καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση. Open the meeting. Like that, can we work according to the... Να εργαστούμε σύμφωνα με την ημερησία διάταξη. Uh, yes, uh, I want to add on this point that έχουμε ένα αίτημα από τον κύριο Πλήτο να βγάλουμε το σημείο 8 από την Ευρωπαϊκή διάταξη, Γενικό Προπολογισμό τη Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2019, όλα τα τμήματα. Γιατί θέλει να καταθέσει εκ νέου τι τροπολογίε ε, τη Επιτροπή μα σε βάση απόφαση των συντονιστών παρά απόφαση τη Επιτροπή ε, και από ό,τι φαίνεται το έγγραφο 6 με όλες τις τροπολογίες που έχουν υιοθετηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και παρουσιάζει μια επισκόπηση της θέσης της Επιτροπής στην πρόταση δεν θα είναι διαθέσιμο πριν το τέλος της εβδομάδας. Από την άλλη, ο κύριος Διντιέ, ο οποίος είναι σκιώδης του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή και ο κύριος Ελίμοβιτς, ο οποίος είναι σκιώδης του ΑΛΔΕ για την έκθεση αυτή, ζήτησαν να διατηρηθεί η ψηφοφορία, να γίνει όπως έχει σχεδιαστεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγώ προτείνω να αποσύρουμε το σημείο από την ημερησία διάταξη. Ενώ αν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα πρότεινα να ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών για να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Ποιος είναι υπέρ να αποσύρουμε το θέμα από την ημερησία διάταξη. Είναι λίγοι οι βουλευτές που είναι εδώ και ποιος θα ήθελε να ρυθμίσουμε το, το ζήτημα. Να ψηφίσουμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν, δύο, ψηφ... ψήφοι ζήτησαν να αποσύρουμε, δύο άτομα να αποσύρουμε και ένας να το διατηρήσουμε. Και καθώς δεν είναι αρκετοί οι βουλευτές, αποφασίζω να αποσύρουμε το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός από Λουγαρικά, φιλάνδικα και κροατικά. Λοιπόν, σημείο 2. Ενημέρωση από τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε, τώρα εργαζόμαστε επί της ε, οδηγίας για την ισορροπία επαγγελματική και ιδιωτική ζωής. Ε, χτες το απόγευμα έλαβε χώρα ο δεύτερος τριμής διάλογος. Ε, συζητήθηκε το θέμα του πεδίου εφαρμογή, καθώς και τα θέματα της γονικής άδεια και της άδειας πατρότητας. Και ενώ η θέση μα είναι πολύ μακριά, ήταν πολύ επικοδομητικές οι συζητήσεις και μπορέσαμε να αρχίσουμε να διερευνούμε διάφορες ε, εναλλακτικέ. Επόμενο τριμερή διάλογο θα λάβει η χώρα στι 6 Νοεμβρίου. Σημείο 3. Μελλοντική τριμερής διάλογη. Έχουμε για τα agencies, για τους οργανισμούς. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε θέμα του αυτού. Επόμενο επόμενος διάλογο θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου το βράδυ, από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 το βράδυ. Point 4. Σημείο 4. Το χρόνο αγόρευσης. Έχουμε μια βεβαρημένη ημερησία διάταξη. Και καθώς είστε πολύ λίγοι, εδώ τώρα αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε σε λίγο πολλούς που θα θέλουν να μιλήσουν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο χρόνος αγορευσής για τους εισηγητές και τους κοιόδης ε, δεν θα είναι πάνω από τρία λεπτά και δύο λεπτά για τους υπόλοιπους βουλευτές. Αλλά θα δούμε. Ίσως ε, όλοι να έχουν αρρωστήσει καθώς δεν έχουν έρθει ακόμη εδώ. Και τότε μπορεί ο καθένα να πάρει το λόγο όσο θέλει. Uh, Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίας της 29 η Αυγούστου. Δεν θέλει κανείς το λόγο γι' αυτό. Επομένως, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στον κύριο Κούκαν, που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ικανοποίηση μου να παρουσιάσω την έκθεση αυτή στους συναδέλφους. Θα ήθελα να τονίσω, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα για το ψήφισμα στην ΑΦΚΟ έχει παραταθεί πολλές φορές από την κυρία Πινέλη, την εισηγήτρια. Επομένως, στο στάδιο αυτό, η κυρία Πινέλη θα παρουσιάσει το τελικό έγγραφο εργασίας αύριο και το σχέδιο ψηφίσματος το 21 Νοεμβρίου καθώς ε, ακόμη δεν είχα το κείμενο της Καθηλιαρμόδιας Επιτροπής, ήταν ε, κάπως πιο δύσκολο να καταρτήσω γνωμοδότηση. Όμως ε, είχαμε πολύ προπερσκευαστική εργασία, προκειμένου να εντοπίσουμε τα κύρια θέματα που διακυβεύονται από τη σκοπιά της δικής μας Επιτροπής. Ε, τεχνικοί περιορισμοί επιβάλλουν το κείμενο να είναι σύντομο, αλλά προσπάθησα να παρουσιάσω κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία από τη Σκοπιά της Επιτροπής Απασχόλησης. Αυτό περιλαμβάνουν μία έκκληση σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για πλήρη σεβασμό με τις κοινωνικές διατάξεις της χάρτας και συστηματική αξιολόγηση επί της συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα τονίζω τη σημασία ότι θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή στα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα. Καλό για αυξημένη ευαισθητοποίηση για τις διατάξεις ε, του χάρτη σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, τονίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται την υποχρέωσή τους σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις ε, του χάρτη και να επιζητούν συμμόρφωση με τα οικονομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελειώνω ημερομηνίε. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα κοινοποιηθείτε εγκαίρως για τις συναντήσεις των σκιωδών. Η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ενυπομονώ να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι γλίτωσε και κάποιο χρόνο για τους μελλοντικού ομιλητές. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σονσάιμερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καλό είναι που εξοικονόμησε χρόνο για υπόλοιπους ομιλητές, γιατί Φαίνεται ότι μαζεύονται πολλοί σήμερα το πρωί που θέλουν ε, κάπως να χωθούν μέσα στη συζήτηση. Να τον συγχαρώ ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω ότι θέσει το σωστό τόνο και για τους υπολείπους. Δεν υπάρχει κάτι τα όσα είπε στο οποίο να μπορώ να, να διαφωνήσω. Το μόνο που έχω να προσθέσω προς ε, μέλη των σοσιαλιστών που ενδεχομένως να σκέφτονται την υποβολή τροπολογιών με βάση το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε. Να ρωτήσω λοιπόν, στις τροπολογίες μας θα μπορούσαμε να τονίσουμε ακόμα περισσότερο ε, τα ζητήματα της Επιτροπής Απασχόλησης, ούτως ώστε όλες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράδειγμα, Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ε, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου, ε, διαφανεί εργασιακέ συνθήκε, δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση. Όλοι αυτοί οι φάκελοι, οι επερχόμενοι, θα πρέπει να τύχουν πολύ διεξοδικού ελέγχου από την ομάδα μα, ούτω ώστε να λαμβάνουν πλήρω υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα ε, στοιχεία του πυλώνα ε, συγγνώμη, της χάρτας των δικαιωμάτων. Αλλά χαίρομαι αυτής εξ αρχής που εργαζόμαστε προς την ε, ίδια κατεύθυνση. Ωραία, κυρία Φεμπέσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Κούκαν, που παρουσίασε τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος. Ήταν πολύ σύντομος και θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει υπό αντίξωες συνθήκες. Πρέπει βέβαια να επιδείξουμε ένα πνεύμα ρεαλισμού και να κατανοήσουμε πραγματικά τον ρόλο μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και να μεριμνήσουμε για τη σωστή εφαρμογή τους ε, στα κράτη-μέλη. Η χάρτα δεν δημιουργήθηκε για να ε, θεμελιώσει νέα δικαιώματα ή να επεκτείνει τα δικαιώματα, απλώς για να γίνουν σεβαστά τα υπάρχοντα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό κατέστα αρκετά σαφές. Αλλά και στο άρθρο 30 είναι σαφές ότι βέβαια τα του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να τα εξετάσουμε ξεχωριστά. Είναι επίση σαφέ ότι η χάρτα δεν επηρεάζει άμεσα τα κρατημέλια, αλλά επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα. Επομένω, επηρεάζει και τα κρατημέλη στο βαθμό που ε, εργάζονται με βάση το πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου. Μετά τη χάρτα πρέπει να τη δούμε ε, συνολικά. Δεν υπάρχει ιεραρχία στα δικαιώματα, κάποια δηλαδή να είναι πιο σημαντικά από άλλα. το Μάιο, μαζί με άλλους εκπροσώπους της Επιτροπής αυτής, ε, επισκέφθηκα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Αυστρία. Και θα ήθελα να μεταφέρω και τη στήριξή μας προς το έργο του οργανισμού. Εντοπίσαμε βέβαια και σημεία βελτίωση ό,τι αφορά την υλοποίηση τη χάρτα. Θα υποβάλω ορισμένε τροπολογίε από αυτή την άποψη και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Όπως είπατε κι εσείς, ε, υποβάλλατε τα πιο σημαντικά στοιχεία από πλευράς Επιτροπής Απασχόλησης. Όπως και όλοι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε ε, από συστηματική άποψη υπόψη ε, τη Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων σε όλα τα βήματα της ε, νομοθετικής διαδικασίας και στην χάραξη πολιτικής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη που προκύπτει από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επομένω, δεν μας απασχολεί μόνο η θέσπιση της νομοθεσίας, αλλά και η εφαρμογή της στην πορεία. Και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σίγουρα μπορεί να είναι σημαντικό σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Σημαντικό εξάλλου είναι να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, συμμορφούνται με τις θεμελιώδεις αρχές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγγράφονται στη συνθήκη. Και έχουμε προσχωρήσει και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα. Συμφωνώ με τη συνάδελφο που είπε ότι δεν υπάρχουν νέα δικαιώματα εδώ και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά ο ρεαλισμό, τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση, ότι όλα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη, δεν είναι μόνο ε, κενό γράμμα. Ο κόσμος να μπορεί να εμπιστεύεται αυτά τα δικαιώματα, να βασίζεται σε αυτά και να έχει τρόπο να δικαιωθεί. Σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Ανθρωπινών Δικαιωμάτων να μην θεωρείται ως μια αρνητική εγγύηση με στόχο να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει, θεωρώ, να προσχωρήσουμε στην άλλη άποψη. Προδραστικά να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει το σωστό πλαίσιο ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ιδίως στον τομέα της απασχόλησης. Είτε έχουμε να κάνουμε το εξάμεινο, είτε με άλλα ζητήματα. Τέλος, η συστηματική προσέγγιση θεωρώ θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και αυτό γενικά είναι εξαιρετικά σημαντικό, πόσο μάλλον τώρα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. κύριο. Σιλικιώτη είναι εδώ ή κάποιο άλλο που εκπροσωπεί την ΓΚΟΕ. No, από την ΓΚΟΕ. Ωραία, ας πάμε στους πρασίνους. Μητροφάνος. Δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω κάποιος άλλος που τον ε, αντικαθιστά. Παρακαλώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι στα όσα ανέφερε ο εισηγητής και οι προηγούμενοι Μιλητέ. Ένα από τα σημεία για εμάς, τα σημαντικά ζητήματα είναι φυσικά και η διαφύλαξη και η εφαρμογή της ομοθεσίας, αλλά και το θέμα της ε, προώθησης ή προαγωγής της κατανόησης και της γνώσης των δικαιωμάτων. Θα υποβάλουμε παντροπολογίες λοιπόν από αυτή την άποψη και να δούμε και πώς ε, θα τα συνδέσουμε όλα αυτά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης γιατί υπάρχει και αυτή ε, η αλληλεπίδραση και με άλλα νομικά εργαλεία που ανέφερε η κυρία Χάρκιν. Πρέπει να γνωρίζουμε και το ρόλο του Equinet σε ό,τι αφορά και την ε, τον σεβασμό προς τα δικαιώματα και την προαγωγή τους, τα οποία συνδέονται και με τα εργασιακά δικαιώματα που μας απασχολούν εμά, αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση ε, στις δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα. Σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Λάμπερτ από το EFTD. Υπάρχει εκπρόσωπος. Όχι. ENF. Κυρία Βεζότο. Παρακαλώ. On this report. Euh, merci, Madame le Président. Okay. Ce sera Dominique Martin. Dominique Martin. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τους προηγούμενους ομιλητές. Ε, να πούμε και εμείς όμως τη δική μας άποψη. Θεωρούμε ότι είναι ε, απλά ένα λογοτεχνικό έργο ε, το οποίο έχει να κάνει ένα προϊόν αμπελοφιλοσοφίας αν θέλετε που μιλάει για την πολιτική ορθότητα ε, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποια σύντομα σχόλια πρωτού συνεχίσουμε. Η κυρία Ινάτ είναι εδώ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάποιος άλλος. from... Όχι, κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, μάλιστα, έχετε το λόγο. Good morning. Καλή σας ημέρα. Ποια ήταν η ερώτησή σας, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, η Πρόεδρος. Θα μπορούσατε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτησή σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. δεν ε, σε ερώτηση. Απλά σας δίνω την ερώτηση, την ευκαιρία ε, να πάρετε το λόγο να προσθέσετε κάτι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την ε, εφαρμογή του χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο λοιπόν, εάν θέλετε να κάνετε κάποια υπόδειξη, κάποια πρόσθεκη, να αναφέρετε κάτι το οποίο απασχόλει ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε σχόλια. Uh, Μάλιστα, το χρονοδιάγραμμα, όπως μας ε, ανέφερε ο κύριος Κούκαν, ε, είναι αυτό που μας ανέφερε. 18 Οκτωβρίου, λοιπόν, η προθεσμία για καταθέση τροπολογιών, 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης 3 ε, Δεκεμβρίου, στην Ολομέλεια ΔΑ. Θα περάσει το Μάρτιο του 2019 το θέμα αυτό. Και έτσι λοιπόν περάσαμε στις ψηφοφορίες. Ας κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα για να βεβαιωθούμε ότι όλοι είμαστε στις θέσεις μας για την ψηφοφορία. Μόνο τρία λεπτά όμως, λέει ο Πρόεδρος. Διαλυματάκι. Uh, this is the first one. Ε, it's this one. Mm. Mr. Κάσα. Ο κ. Κάσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και πρωτού ψηφίσουμε, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα μόνο. Όπως θα ξέρετε, δολοφονήθηκε ένα δημοσιογράφο στη Βουλγαρία. Δεν ξέρουμε ακριβώ τα αίτια. Τρίτο φέτο ε, στη Μάλτα, στη Σλοβακία. Τώρα και στη Βουλγαρία. Πρόκειται και για εργαζόμενου, πέρα από το γεγονό ότι είναι δημοσιογράφοι δηλαδή. Θα πρότεινα ενό λεπτού σιγή για να τιμήσουμε το έργο των ε, δημοσιογράφων αυτών, οι οποίοι τυχαία ερευνούσαν ε, θέματα ε, διαφθορά. Ενό λεπτού σιγή λοιπόν προτείνω, λέει ο κύριο Κάζα, προ τιμή τη δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε. Δεν βλέπω κανένα να ενίσταται, λέει η πρόεδρος, οπότε και θα κάνουμε ενός λεπτού σιγή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την επιστολή. Μία γνωμοδότηση για την κινητοποίηση του Ταμείου EGF. Υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία, ναι, συγγνώμη. And the vote is closed. Και πέρασε. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έκθεση Hetman για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ. και κατόπιν αιτήματος της ομάδος της ΓΚΟΕ, οι 65 και 144 τροπολογίες θα ψηφιστούν ως προσθήκες στο συμβιβασμό 11 και στο συμβιβασμό 22. Και να ξεκινήσουμε. Δεν έχω την κάρτα για να ψηφίσω, λέει η Πρόεδρος. Θα δω πώς θα τα βγάλω πέρα. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 61. Έναρξη ψηφοφορίας. Και πέρας. Απορρίπτεται. 20 ψήφοι υπέρ και 20 κατά ισοψηφία. Η δική μου κάρτα έκανε τη διαφορά, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Έλεγχος ζητείτε. Ηλεκτρονικά έχουμε και την 62. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Σχολέκτος μικροφώνου. Προχωράμε με τη συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το 65, το οποίο το ψηφίζουμε ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ωστόσο την 65. Ψηφίζουμε παρακαλώ την 65. Πέρας απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Και προχωράμε. 68 και 69. Ταυτόσιμες. 68-69 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία Συγγνώμη, τη συμβιβαστική, λέει η πρόεδρο. Όχι, την τροπολογία, 70. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 είναι η ψήφη κατά, 18 υπέρ. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 σε τμήματα. Πρώτο το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Και έτσι περνάμε στην συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. 14 υπέρ. Να ξαναδούμε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Α, συγγνώμη. Πάμε κατευθείαν στην 98. Καταπίπτουν τα υπόλοιπα τμήματα. Ψηφίζουμε την 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99, δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 ψήφοι υπέρ. 14 της Επιτροπής Πολιτισμού δεν ψηφίζουμε. Η 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 108 108 ναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 λοιπόν, ναι. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 125 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Θα έλεγα, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 125 να είμαστε σίγουροι ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 127 ε, υπέρ. Έλεγχος για την 126 παρακαλώ ηλεκτρονικά έλεγχουμε. Ψηφίζουμε για την 126. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Πα, ξανά για την 20 παρακαλώ ψήφισμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η δύο του πολιτισμού, έτσι επιτρέπει πολιτισμού σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έκτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η πέντε του Επιτροπής Πολιτισμού, όχι. Ναι, ναι, ναι, η πέντε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η έξι της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η επτά, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 11 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 17 της Επιτροπής Πολιτισμού πάντα. Ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Η 18 δεν ψηφίζεται, 20 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 20 της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται τρεις ψήφοι διαφορά. 21 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος και για την 21 τη Επιτροπή Πολιτισμού και ψηφίζουμε παρακαλώ. Και πέρασε. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε για την 144 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 144. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 ψήφοι κατά. 18 υπέρ. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 καταπίπτει. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στο 1 των τελικών σκέψεων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές απορριπτωτικά. 1α ή 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο 1β παρακαλώ η τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Στα υπόψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 8. Ψηφίζουμε. Και πέρασε. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε παρακαλώ τη 10. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στις συλλογικές σκέψεις. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4 της Επιτροπής Πολιτισμού καταπίπτει. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 31 της κυρίας Τραμπέσιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 27 η ψήφη υπέρ. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ταυτόσιμες οι τροπολογίες 51 και 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε 30 ψήφοι υπέρ, 8 ψήφοι κατά, 4 αποχές. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή. Και να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη έκθεση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. The interim report. Ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να ψηφίσουμε την ε, απόφαση ε, που πήρατε να αφαιρέσουμε την ύψη διάταξη το σημείο 8. Εγώ νομίζω ότι σε μια δημοκρατία κάθε φορά το ίδιο πρέπει να γίνεται. Την τελευταία φορά για την απόσπαση των εργαζομένων διατηρήσαμε την απόφαση να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα αλλάξαμε και περάσαμε ε, να ψηφίσουμε μόνο στους συντονιστές. Έτσι λοιπόν θα σας παρακαλούσα αν, να θέσουμε σε ψηφοφορία το αν θέλουμε να διατηρήσουμε στην ημερή της αδιάταξης το σημείο 8 όσο έχει. Let's vote on item 7 first and then... Να ψηφίσουμε πρώτα για το 7 και θα επανέλθουμε για το 8. Yes, but the point of order is... Κοιτάξτε το διαδικαστικό όμως το έθεσα. Απλώς θέλω να το κάνω εγκαίρος. Μετά το σημείο 7. Έθεσα το διαδικαστικό θέμα μου και τι προτείνω. Μάλιστα. Αλλά θα ψηφίσουμε πρώτα για το 7. We stop by voting on amendment. Περνάμε στην τροπολογία 4 για το σχέδιο γνωμοδότησης, ενδιάμεση έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, υπορρίπτεται. Τροπολογία 6, έχουμε προφορική Τροπολογία από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 24 ψήφους κατά. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11, 12, 13 έχουν αποσυρθεί. Πάμε στη 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε 16, 17, 18, 19, 21 και 20 που αποσύρονται Επομένω, πάμε στο κτιμώντα τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε το εκτιμώντα C. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται για μία ψήφο. Πάμε στην τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε Προφορική τροπολογία από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, για την τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο σημείο 8. 20 προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό Έτο 2019. κύριε Σπριέτο. Θέλετε το λόγο, κύριε Πριέτο. Δεν είναι εδώ. Θέλει να καταθέσει εκ νέου τις τροπολογίες της ΕΜΠΛ βάσει απόφασης των συντονιστών παρά απόφασης της Επιτροπής. Και από την άλλη, ο κύριος Διντιέ και ο κύριος Καλβιασαμπών ζήτησαν ε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όπως έχει σχεδιαστεί. Παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Γιονγκέριους. Κύριος Κάνσα. Κύριε Γιονγκέριους καταρχήν. Εγώ κατάλαβα στην άνοιξη αυτή τη συνεδρίαση είχατε ήδη ψηφίσει στο να αφαιρεθεί από την ημερική διάταξη αυτό το σημείο. Αυτό κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, ε, γιατί καταρχήν αποφάσισε η Επιτροπή να αφαιρέσει το σημείο αυτό και τώρα επανέρχεται. εγώ εκ μέρους και του συναδέλφου θεωρήσαμε το εξή. Καθώς δεν υπάρχει απόφαση των συντονιστών να κατατεθούν εκ νέου αυτές οι τροπολογίες και δεν βλέπουμε την ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να μείνουμε στην απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή πριν έρθει ο κύριος Σαμπόρ στην αίθουσα. Δηλαδή να μην ψηφίσουμε επί της πρότασης αυτής. να το αφήσουμε όσο έχει. Κύριος Κάσα. Τον έφερε συνάδελφος. Είχαμε τρεις βουλευτές μόνο παρόντες ε, όταν ψηφίσαμε και αποφασίσαμε στην αρχή της συνεδρίασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του κυρίου Καλβέσαμον και του κυρίου Ντιτιά και θέλουμε να γίνει ψηφοφορία σήμερα. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ως ένας άνθρωπος που ήμουν εδώ, στην αρχή της συνεδρίσης και όντως ψηφίσαμε, να πω ότι τι συνέβη. Όντως ψηφίσαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ε, όσοι ήταν εδώ, εγκαίρως, εγώ ήμουν άλλοι δεν είσαστε. Και η πρόεδρος είπε τότε, καθώς ε, δεν υπάρχουν πολλοί εδώ, αλλά οι, δύο, ε, οι τρεις που ήταν ψήφισαν δύο προς ένα νομίζω για την αναβολή. Και είπατε, αποφασίζω να αποσύρω το σημείο αυτό. Νομίζω ότι ναι, θα μελιώδες ότι όσοι εμφανίζονται συνεδριάσεις και ψηφίζουν, αν ε, ανατρέπονται οι διαδικασίες επειδή οι υπόλοιποι έρχονται 20 λεπτά μετά και δεν ήταν εδώ. Δεν ε, είναι ουσιαστικά σοβαρός τρόπος εργασίας για ένα σοβαρό κοινοβούλιο. Κύριε Μακιντάρ, εγώ υποστηρίζω τον κύριο Καλβεσαμπών. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συνεκτικοί. Ή θα αποφασίσουμε αν θα καταθέσουμε γνώμη τη τροπολογία ή όχι και νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε καταθέσει εκ νέου τροπολογίες, δεν το αφήσαμε στους συντονιστέ να το αποφασίσουν και νομίζω ότι προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη δημοκρατία θα πρέπει να ψηφίσει η Επιτροπή μας. Κάσα. Κύριος Κάσα, πέρα από το γεγονό ότι έχουμε διαδικαστικούς κανόνες, ίσως ε, μπορεί να μας πει η γραμματεία ότι υπήρχε απαρτία σήμερα όταν ελήφθη απόφαση. Ε, Παρακαλώ. Να πω ότι δεν πίστευα ότι υπήρχε απαρτία και γι' αυτό η πρόεδρος τη στιγμή της συνεδρίασης είπατε, πρόεδρε εσείς, καθώς δεν είναι αρκετά άτομα εδώ, αλλά όσοι είναι ψήφισαν δύο προς ένα, εγώ ως πρόεδρος αποφασίζω να αποσύρω το σημείο, αυτό, είπε. αυτό είπατε. Αυτό που λέμε είναι ότι στα διαδικαστικά της συνεδρίασης ε, έλαβε χώρα ψηφοφορία όταν έπρεπε και εσείς αποφασίσατε να αποσύρετε ε, το σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται διαδικαστικά ή όχι, αλλά αυτό συνέβη. well, those who are really formal guys, like this one. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι που είναι τυπικοί, όπως ε, εδώ ο συνάδελφος, είναι ξεκάθαρος. Είναι οριστική έγκριση της ημέρησης διάκριση και εγκρίναμε την ημέρηση διάταξη όταν ξεκίνησαμε τις συνεδρίες. Λέγοντας ότι θα αποσύρουμε το σημείο αυτό από την ημέρηση διάταξη. Εγώ είμαι πρώην υπουργό πολιτισμού και ξέρω ότι και το χάος μπορεί να οδηγήσει σε φανταστικά πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν η πλειονότητα των μελών αυτής της Επιτροπής ε, προτιμά το χάος, κύριε Κάσα. Ναι, καταλαβαίνω την κατάσταση, τι συνέβη σήμερα το πρωί, αλλά τώρα έχουμε πλειοψηφία των μελών. Ζητάμε μια ψηφοφορία για το αν θα ψηφίσουμε για αυτό το συγκεκριμένο φάκελο ή όχι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψετε στα μέλη να αποφασίσουν αν μπορούμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Κύριε Γιονγκέριος, για τη σαφήνεια των εργασιών μας δεν μπορούμε να αλλάζουμε την ημερησία διάταξη κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχει δίκιο η γραμματεία. Έχει βγει το θέμα με την ημερησία διάταξη. Δεύτερον. Αλλά αυτό για να απαντήσω στο σχόλιο της κυρίας Μάκεντάιρ. Στο προηγούμενο έτος, τους συντονιστές αποφασίσαμε για το αν θα καταθέσουμε ή όχι εκ νέου τροπολογίες και όχι στην Επιτροπή. Δεν συνέβη αυτό εδώ και μας ε, εξέπληξε ότι είναι στην ημερησία διάταξη χωρίς ε, απόφαση των συντονιστών να προχωρήσει. Για να είμαι σαφής, θέλω να ενταχθώ σε αυτό που ανέφερε η κυρία Μακεντέρ. Κοιτάξτε, de Εντάξει, η δημοκρατία συνίσταται να δίνετε το λόγο, το υπερθυμίζω. Ο κύριο ε, Πριέντο θέλει να καταθέσει εκ νέου τη τροπολογίες Επιτροπή Επισχόλησης βάσει απόφαση των συντονιστών παρά απόφαση της Επιτροπής και ε, ότι το έγγραφο 6 με όλες τις τροπολογίες που έχουν υιοθετηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και δίνει την επισκόπηση της Επιτροπής για την προτεραιόμενη απόφαση ως έχει δεν θα είναι διαθέσιμο πριν το τέλος αυτής της εβδομάδας. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η δική μου πρόταση εξακολουθεί να είναι ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε το θέμα με την ημερησία διάταξη. Καθώς αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα. Και ελπίζω να μπορείτε να το δεκτείτε. Κύριε Σμάν. Κυρία Πρόεδρε, ενημερώθηκα ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης, μάλλον από ό,τι ξέρω, έχουμε γενικά μεγάλη συμφωνία και νομίζω ότι συμφωνούμε ιδιαίτερα ω προ τα διαδικαστικά. Η Άκνε δίκιο έχει ότι καλύτερα θα ήταν να το έχουν αποφασίσει αυτό οι συντονιστέ. Δεν έγινε αυτό. Στην ψηφοφορία ήμουν ε, εκεί. Ήμουν η μία ψήφο κατά. Αλλά όταν το ψήφισαν υπέρ, ε, οι υπόλοιποι τι να κάνουμε, 30. Δεν το κάνουμε για να αναβάλουμε ψηφοφορίες, αλλά για να πούμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί πάντα στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης ήμασταν προσανατολισμένοι στο πώς θα βρούμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Πόση ώρα θα πρέπει να κρατάω το χέρι μου ψηλά. Α, μάλιστα, ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που υπήρχε στον κόσμο του οικονομολόγου. Γιατί ό,τι και να υπήρχε, υπήρχε το χάος. Εγώ είμαι λοιπόν ειδικό, αλλά απέναντι στο χάος υπάρχει κοινή λογική και δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, να υποστηρίζει κανείς ότι μία ψηφορία δύο προς ένα ε, καθορίζει μία συνέλευση ε, τελικά θα πρέπει να φτάνουν όλοι 9 παρα 10 δευτερόλεπτα για να χειραγούν του υπόλοιπου. Αυτό που ζητώ δεν είναι ε, ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Ε, πλώς ζητώ να υποβάλουμε μία απόφαση τέτοιας κατηγορίας που ε, εδώ διακυβεύει όχι μόνο τις τροπολογίες ε, του Σέργιο αλλά και τη δημοκρατική διαδικασία. Ζητώ ουσιαστικά να λάβουμε μία απόφαση με απαρτία. Απλώς αυτό. Νομίζω ότι εξαρτάται και από την ε, ευφυΐα και την ευελιξία του Προεδρείου και της Γραμματείας να εκτιμήσει ότι καθώς δεν υπήρχε η απαρτία στην αρχή θα ήταν πολύ πιο δημοκρατικό αν αποφασίζαμε όσοι είμαστε εδώ. Αλλά οι τρεις ε, που ήταν στην αρχή για μια τέτοια κατηγορία, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να παρέμβει η κοινή λογική. Χωρίς ε, τώρα εδώ να είμαι κανονιστικός. Ευχαριστώ, κύριε Λαβριλέ. Πρόεδρε, και εγώ ήρθα στι 9.30, αντί να έρθω στι 9. Βέβαια, εντάξει, είμαι ένοχο, καθυστέρησα μισή ώρα. Εγώ είδα την ημερησία διάταξη πριν έρθω. Στην ημερησία διάταξη λέει έγκριση τη ημερησία διάταξη. Είναι το σημείο 1. Και η ημερησία διάταξη είναι από τα σημεία 2 μέχρι το σημείο 8. Και στην ουσία διάταξη πουθενά δεν λέει ότι θα προτείναμε σε ψηφοφορία στις 9 ότι θα αποσυρώταν το σημείο 8. Αν λεγόταν ότι υπήρχε μια πρόταση απόσυρση του σημείου 8, θα είχα φτάσει στις 9 αντί να φύγω στις 6, θα έφυγα στις 5 από το σπίτι μου για να αποφύγω και το ποδηλιάρισμα στην ίσοδο των Βρυξελών, ήρθα να συμμετέχω σε αυτή την ψηφοφορία. η ψηφοφορία όταν έχουμε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι θα έχουμε ψηφοφορία και μάλιστα δεν είναι και ίσονο σημασία. Αν δηλαδή είχατε γράψει μέσα η διάταξη ότι θα είχαμε μια ψηφοφορία για να αποφασίσουμε αν θα διατηρήσουμε, θα αφαιρέσουμε το σημείο αυτό από την ημερησία διάταξη, θα είχα έρθει. Η έγκριση ημερησία διάταξη εδώ και τέσσερα χρόνια κρατάει τρία δευτερόλεπτα. Γιατί ουσιαστικά η ημερήσια διάταξη τη Επιτροπή είναι αυτά που αναγράφεται στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, όπω ζήτησε και ο κύριο Σαμπόν, θα έλεγα να προχωρήσουμε ή να ψηφίσουμε για το σημείο 8, γιατί εγώ ήρθα και το σημείο 8 ήταν γεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Ποτέ δεν λέγατε ότι θα ψηφίζαμε για την ενδεχόμενη απόσυρση του σημείου 8. Μου φαίνεται λογικό λοιπόν. I'm not sure I understood everything, but there Δεν είμαι σίγουρη ότι τα κατάλαβα όλα. Δεν υπήρξαν όμως σχέδια προξικοποίηματος. Θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτά που είχαμε στην ημερησία διάταξή μας και να είμαστε στον έτον πιο αποτελεσματικοί. Δώστε μου λίγα λεπτά με τη γραμματεία και θα βρούμε λύση. Just sit and relax. Don't leave the room. Καθίστε και χαλαρώστε, μην, μην αποχωρήσετε από την αίθουσα, γιατί τότε μάλλον θα έχουμε πάλι πρόβλημα. take seats. Καθίστε, αγαπητοί φίλοι. We will uh, Θα ψηφίσουμε, αλλά καταρχήν θα δώσω δύο λεπτά στη γραμματεία. Έχετε το λόγο. Αν μου επιτρέπετε είναι όπως στην Ολομέλεια. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη στην έναρξη της συνεδρίασης από όσους είναι παρόντες. Εν συντομία, αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Ήταν στην ημερήσια διάταξη ο γενικός προπολογισμό. Και μάλιστα υπήρξε και ένα μήνυμα ότι θα ξεκινήσουμε στις 9, έτσι, δεν υπήρξε κάποια απάτη εδώ. Τώρα να ψηφίσουμε, εντάξει, γιατί αυτό θέλετε. Τουλάχιστον όσο το ζητήσατε. I understand that it will be seen upon ε, ε, ε, in a way that I don't want it to, to... Αν δεν ψηφίσουμε, μάλλον θα δημιουργηθούν κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις. Ας ψηφίσουμε επομένω. ας περάσουμε για τη διαδικασία. Μίστε Mr. Je... Ακριβώς αυτό ήθελα και αυτό σας τιμά, κυρία Πρόεδρε πέραν των τυπικών στοιχείων υπάρχει και το δημοκρατικό αίσθημα και σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Σας θυμάμαι πραγματικά. Mr. Sean Simon. Κύριε Σάιμον, να πω μόνο ότι αν χάσουμε την ψηφοφορία μπορούμε να την ξανακάνουμε μετά που θα είναι άλλοι συσχετισμοί. Who knows, who knows. Ποιος ξέρει. Start with this, uh, and we vote on uh, employment. Ξεκινάμε λοιπόν. Put the item to the vote. We vote if they want yeah. to vote on yeah. it. Yes, we start by voting on. Shall we vote on this? Πρώτα θα ψηφίσουμε για να δούμε αν θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. We check it to be really... Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. No, no, no. the vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την 5503 ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, λέω. 5504 της απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 5505. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5506. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5508. Της απασχόληση υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 5508. Πέρασε. 30. Απορρίπτεται. Πέντε πέντε δέκα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 5510. And the vote is now closed. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. 55-11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Are you doing something with your hands that is the other way around? Shall we use uh, the buttons through all the voting because some of you are showing in a different way. Ας ελέγχουμε ηλεκτρονικά όλες τις ψηφοφορίες γιατί μπερδευόμαστε. 55-11 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται με 32 ψήφους κατά. 55-13. Άρχεται. And the vote is now closed. Πέρασε. And 32 on Rejection. Απορρίπτεται. 55-14. Άρχεται. 5-14. And the vote 31 against and 1 in favor. Απορρίπτεται. 55-17. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now closed and it's... Πέρας. Απορρίπτεται. Four in favor. Employment 55, uh, 18. 55-18. Άρχεται. And the vote is now closed and it's Πέρας. Απορρίπτεται. 55-19. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 55-21 της απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55-43 και 55-44 αυτές οι δύο απορρίπτονται. Όχι, όχι, Τις ψηφίζουμε από κοινού. «5543» και «5544» ψηφοφορία από κοινού άρχεται. And 29 in favor and Εγκρίνονται. 55-27 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55-31. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται.

Άρχεται. Έγκρινεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν. That we proceed. Yeah. Well, it's, we seem to be rather Um, unified uh, through this uh, voting uh, result. Τουλάχιστον είμαστε ενωμένοι σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη μέσα διάταξη. Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση των ναυτικών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Σύντομα. Από τις Κανάριες νήσους. Τις Αζόρες μάλλον. Some order oh. Η κυρία Ριμπέριο θα περιμένω κυρία Πρόεδρε για να υπάρξει ησυχία στην αίθουσα. Ωραία, θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια για το σημείο 9, ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση των ναυτικών. Η κυρία Ριμπέιρο κατάγεται από τις Αζόρες, επομένως ε, τα ξέρει αυτά τα ζητήματα και πρακτικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για τη συμπατική αναφορά που κάνατε στις Αζόρες η αυτόνομη περιοχή της, ε, των Αζωρών ε, είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα και φυσικά τα θέματα αυτά απασχολούν τους Πορτογάλους και τους κατοίκους των νήσων. Η βελτίωση της εκπαίδευσης βρίσκεται στην κορφή των προτεραιοτήτων μας ε, το να δώσουμε ικανότητες και δεξιότητες στους πολίτες μας αφορά πολλού πολλούς και φυσικά δεν είναι εξαίρεση ο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ξέρουμε ότι με τη θαλάσσια οδό κινείται το 90% των εμπορευμάτων, με το εξωτερικό και το 40% των εμπορευμάτων σε εσωτερικές οδούς και υπάρχει τεράστιος οικονομικός αντίκτυπος και στη δημιουργία θέσεων εργασία. Ξέρουμε ότι στον τομέα αυτό το να εγγυηθούμε την επιστοποίηση πίση την εξειδίκευση και την κατάρτιση των ναυτικών προκειμένου να μειώσουμε τις απειλές ε, κατά των ανθρώπινων ε, ζωών και των αγαθών ε, στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επί των σκαφών είναι πολύ σημαντικό, είναι απαραίτητο λοιπόν ε, να θέσουμε ελάχιστα επίπεδα κατάρτισης και ελάχιστες απαιτήσει για την εργασία και την ασφάλεια επί του σκάφους. Επίσης, καθώς ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών είναι παγκοσμιοποιημένο, πρέπει αυτές να συνάδουν με τις διεθνείς συμβάσεις και να προσαρμοστούν στις πρόσφατες εξελίξεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την αναθεώρηση αυτής της οδηγία σε σχέση με το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης των ναυτικών που καταργεί την προηγούμενη ε, οδηγία του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναδιατυπώσει και να πλουστεύσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να καλύψει τα κενά που έχουν ήδη εντοπιστεί ε, καθώς οι ναυτικοί αλλά και όσοι προέρχονται από τρίτες χώρες να εργάζονται σε συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν θέλουμε να εγγυθούμε την ασφάλεια και την ισότητα στις θέσεις εργασίας χωρίς να ξεχνάμε την προστασία των ναυτικών ω εργαζόμενοι. Αυτό αυτού πρέπει να είναι η δική μας ανησυχία ως Επιτροπή απασχόληση και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, για τους εργαζόμενους, είτε σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση ευκαιριών εργασίας στα κράτη-μέλη, είτε σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των προσωρινών πιστοποιητικών. Όλη αυτή η διαδικασία αναγνώρισης ε, των πιστοποιητικών, ε, των αυτών που προέρχονται και από τρίτες χώρες, θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύπλοκη διαδικασία με το REFIT, που ενέχει μια σειρά διπλωματικών μηχανισμών και αυτό χωρίς ε, να μιλάμε για άλλα μέτρα που μπορεί να εφαρμοστούν. Επομένως, η οδό θα πρέπει να είναι να πλουστεύσουμε τη διαδικασία και να την ψηφοποιήσουμε και να εγγυηθούμε ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν όλα αυτά και όχι να ε, επιτείνουμε τις προθεσμίες, να παρατείνουμε τις προθεσμίες. Ε, ε, ουσιαστικά θα πρέπει να σεβεστούμε ε, και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις καθώς και τις αρχές της επικουρικότητας. Εγώ κατανοώ πρέπει να ακολουθήσουμε μία οδό σύγκληση προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και όταν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ε, πολύπλοκες ε, διαδικασίες από τα κράτη-μέλη, ενώ μπορεί με εύκολο τρόπο να λυθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ουσιαστικά αυτή την οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα να πω ότι στην τροπολογία μου υπαριθμών 3 ε, έχω βρει κάποια λάθη στη μετάφραση στην αγγλική εκδοχή που αλλοιώνουν εντελώς την πρότασή μου. Η τροπολογία μου λέει το εξή και θα την αναφέρω. Ε, πέραν αυτού, αυτή η ναυτική θα πρέπει να είναι στόχος αξιολόγησης από την πλευρά των κρατών μελών και αν είναι απαραίτητο να ε, δεχτούν για κατάρτιση, τέλος της παράθεσης. Και επομένως ε, θα ήθελα να γίνει η κατάλληλη διόρθωση στη μετάφραση της τροπολογίας υπαριθμών 3, προκειμένου να έχουμε πρόβλημα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. τον αυτό, Πρόεδρε, να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω ε, την άποψη των συναδέλφων και φυσικά θα λάβω υπόψη τα σχολιά τους προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε μια καλή συμβαστική πρόταση. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ριπέρου, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή αυτή και παρακαλώ στις παρεμβάσεις σας να περιοριστείτε στα δύο λεπτά αγαπητοί συνάδελφοι. Το λόγο έχει ο κύριος Πάντρας, κοιόδης εισηγητής. Έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς ο μιλητής. Σα ευχαριστώ. Είχα την χαρά και την τιμή να εργαστώ για μια ναυτιλιακή επιτρία χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η εκπαίδευση των ναυτικών να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε απόκληση από τα πρότυπα αυτά και μόνο και μόνο επειδή καθυστερούμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προδιαγραφών εμεί. Θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα εφαρμόσουμε τι προδιαγραφέ. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή. Είναι επίση σημαντικό τα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούνται προ την κατεύθυνση αυτή. Σε μια κατάσταση όπου είναι λίγοι οι ναυτικοί από τι τρίτε χώρε. Άρα δεν ε, είναι ενδεχομένω η ενδεδεγμένη λύση των να τα κονδύλια προ την ε, επαλήθευση των ικανοτήτων αυτών. Θα πρέπει να επιτρέπεται λοιπόν αυτή η απόκληση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι υψηλέ οι ικανότητε και οι προδιαγραφέ που ακολουθούνται στην εκπαίδευση των ε, ναυτικών μα, ό,τι αφορά για παράδειγμα τα ψηφιακά μέσα, προκειμένου να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Ριπέιρο για τη δουλειά που έκανε αλλά έχουμε κάποια θέματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν και σίγουρα θα τα θίξουμε αυτά στη συνάντηση των σκιωδών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις σχετικές προθεσμίες. Και θα ήθελα να, κατα... να υποβάλω και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά αναμένω ότι η συνεργασία θα είναι άριστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην Γιάννα Τούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι περίεργο που δύο από τους έξι ε, βουλευτές είναι οι ίδιοι σκιώδεις. Ε. Μου, θυμά, μου θυμίζει κάτι που είχε γράψει ο Hemingway, ότι σε κάθε λιμάνι μπορεί να συναντήσει κανείς από έναν ε, μεθυσμένο εστονό. Τα πράγματα περιπλέκονται σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι πολύ τεχνικό ο χαρακτήρα και προφανώ αυτό επηρεάζει τι συνθήκε εργασία των ναυτικών και έχει ζητηθεί η ε, η υιοθέτηση των προδιαγραφών αυτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας. Ως κοιότης, λοιπόν, θα ακολουθήσω τη γραμμή του Άλντε. Εκφράζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς αντίθετες απόψεις σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά και το κοινωνικό dumping, οι πλήκτητε μιλάνε για διακύβευση του μέλλοντος της ελληνικής της ευρωπαϊκής ναυτιλίας δεδομένων των υψηλών προδιαγραφών και είναι δύσκολο όταν υπάρχει απόπειρα να βγουν εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας τα πλοία. Η προθεσμία για τις τροπολογίες αναφέρθηκε ήδη από την εισηγήτρια. Θα καταθέσουμε λοιπόν και εμείς τροπολογίες όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος η Ιαρίκ δεν είναι εδώ. Τον αντικαθιστά κάποιος. Όχι. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην κυρία Καρίμα Ντέλη. Είναι εδώ. Όχι. Δεν προσωπεί κάποιος άλλο τους πράσινους. Όχι. Ο κύριος Γκέρι και αυτό δεν θέλει το λόγο. Η κυρία για να του μίλησε No is here representing EFDD. Από το EFDD είναι κανείς. Ο κύριος Μαρτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Ριμπέρο για την έκθεση για τις ελάχιστες προδιαγραφές των ναυτικών. Έχετε δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αποτελεσματική σε αυτή την διαδικασία επαλήθευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θέλει να δώσει τρία χρόνια στις ξένες χώρες για την ε, εκπαίδευση των ναυτικών είναι πολλά. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε την ασφάλεια των ναυτιλωμένων, γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Σύμφωνα με λοιπόν μαζί σας και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι απαράδεκτο να μα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδηγία αυτή, την προτοσία αυτή η οδηγία, χωρί την εκτύπου σε ό,τι αφορά και τον αντίκτυπο που θα έχει στου Ευρωπαίου ναυτικού. Παρά το γεγονό ότι γράφει, θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία για του ναυτικού. Στην σελίδα 4 αναφέρει και παραθέτω ότι η διαδικασία δεν λαμβάνει υπόψη είναι τον αριθμό των καπετάνιων και ναυτιλωμένων που ενδεχομένως θα α, τους προσλάβουν και θα τους απασχολούν από αλλοδαπές τρίτες χώρες και είναι την παράθεση εδώ γιατί φαίνεται ότι αυτό δεν ανησυχεί κανέναν στην Ευρώπη ότι αυτοί που προσφέρουν δηλαδή θέσεις εργασίας. Καταθέσαμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Και έτσι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, επαναλαμβάνω, είναι η 16 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, στις 26-27 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης στις 22 Ιανουαρίου του χρόνου. Σας ευχαριστώ και έτσι περνάμε στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στο λόγο θα έχει η κυρία Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Σκιωδούς εισηγητή για μια καθυστέρηση, για μια αναβολή της προθεσμίας. Όπως ξέρετε υπέστη μια κύρωση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε κάποιες επίσημες συνεδριάσεις και βλέπω ότι ο συνάδελφος Κλοκλορόλα Μηδιά, γιατί και αυτό επλήχθη από την κύριο Ζητώ συγγνώμη λοιπόν προ του σκιώδει εισηγητέ. Ε, υπεστήσαμε κυρώσει, αλλά ήταν για καλό σκοπό, για ευγενή σκοπό, για να προασπιστούμε τα συμφέροντα των ερμηνέων. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Προσαρμογή στην Καμπακοσμιοποίηση, λάβαμε βάση τη πρόταση την οποία και υπέβαλα Λάβαμε 76 τροπολογίες ε, για την πρόταση αυτή. Καταφέραμε να συνάψουμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αιτιολογικών σκέψεων της έκθεσης. Ε, και από 10 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε λοιπόν τι εργασίε για το κομμάτι αυτό. Σε ό,τι αφορά τι συνεδριάσει των σκιωδών τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί προφανώ και ε, τρέχει ο χρόνο και έχει σημασία ο χρόνο ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή ω κοινοβούλιο τουλάχιστον. Θέλουμε μέχρι τον Νοέμβριο να έχουμε δώσει σαφεί κατευθυντήριε γραμμέ σε ό,τι αφορά και το Συμβούλιο και σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν τρεις ε, συναντήσεις 23 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου και 13 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης προβλέπεται για τις 19 ή 20 Νοεμβρίου και ως εκ τούτου Δεδομένων και των τροπολογιών ε, που έχουμε λάβει, θα είναι πάρα πολύ επικοδομητική η εργασία που έχουμε μπροστά μα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή. Όπω σα είπα, πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και αναγκαίο για του εργαζομένου και θα πρέπει να το με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο σε ό,τι αφορά την ένταξη των ατόμων αυτών που έχουν χάσει τη δουλειά τους σε νέες θέσεις απασχόλησης να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής και τους βοηθούς τους να παρευρεθούν στην συνάντηση που θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα σε ό,τι αφορά το έργο Caterpillar στο Σαρλερούα, το οποίο αποτέλεσε ένα έργο ε, ε, με τα ρύθμιση Ford Gang σε ό,τι αφορά το τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία θα μα επιτρέψει να εξηγήσουμε με ένα συμπληρωματικό τρόπο πώ μπορεί να υπάρξει αυτή η αλλαγή θέσει απασχόληση σε περιοχέ που έχουν υποστεί μεγάλου κλειδονισμού, μεγάλα σοκ, γιατί έχει κλείσει μια μεγάλη εταιρεία. Πώ μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ότι εργαζόμαστε όχι μόνο σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου, αλλά ότι δίνουμε και δείχνουμε σε όλα τα επίπεδα, στους ακαδημαϊκούς, στις κοινωνίες, πώς πρέπει να οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο η κοινωνία μετά από τέτοιες μεγάλες ε, αλλαγές, για να μην υπάρχει ουσιαστικά απερίμωση ολόκληρων περιοχών σε περίπτωση που κλείνουν κάποιες μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες. Σας καλώ λοιπόν από 12.30 και μετά ASP 3 και δεν έχω και τα γυαλιά μου να δω την αίθουσα να τη διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς που θα λάβει χώρα αυτή η εκδήλωση στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα. Σας ευχαριστώ, λέγει Πρόεδρος, κύριε Αρένα. Το λέγω να πάρει ο κ. Παντεκάντελάρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, συνάδελφοι. Ε, πράγματι, όπως ε, αναφέρει και η συγγήτρια, ε, αρκετές ε, συνεδριάσεις των σκιωδών δεν έγιναν. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τι ταχύτητέ μα τι επόμενε εβδομάδε. Χθε το βράδυ έγινε μια πρόταση, λάβαμε την πρόταση μάλλον συμβιβασμού για τα εκτιμώντα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, αλλά να τονίσω ότι ακόμα θα πρέπει να υπάρξουν προσαρμογέ. Όπω θα θυμάστε, το ίμιση των τροπολογιών του προσχεδίου ε, μιλούσε για μία τροποποίηση του τίτλου. Και εγώ δεν λέω ευθύ εξ αρχή όχι στην αλλαγή του τίτλου, αλλά για το ΕΛΚ αυτό δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι θέμα ουσία. Το θέμα ουσία είναι η προσβασιμότητα και ο σκοπό του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Για την πρόσβαση, μπορώ να σα πω ότι μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει ε, συνένεση να γίνει πιο προσβάσιμο το Ταμείο, ε, μειώνοντα τον το κατόφλι του αριθμού των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα σημείο κίνηση. Δεύτερον, σε ό,τι φορά το σκοπό, στο άρθρο 3 τη πρόταση τονίζεται ότι πρέπει να έχουμε ένα απρόοπτο συμβάν για την ε, ε, διοχέτευση των ε, κονδυλίων. Είναι λοιπόν ένα ταμείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από τις απολύσεις σε αντίθεση με τα διαφορετικά ταμεία. Είναι σαφής η διαφορά. Αυτή η αρχή επιβεβαιώθηκε και στην πρώτη συζήτηση που κάνουμε για αυτό το ταμείο, αλλά βλέπω από την, ε, τις συμβαστικές προτάσεις ότι αυτό θα μπορούσαν να διατυπωθεί ακόμα πιο σαφώ για να μην υπάρχει καμία πολιτική παρανόηση και παρερμηνία. Πραγματικά προσβλέπω στι συνεδριάσει των ε, σκιωδών που ελπίζω να λάβουν χώρα η μία μετά την άλλη και έτσι να υπάρξουν και συμβαστικέ προτάσει για τι τροπολογίε. Ευχαριστώ. Thank you. I'll give the floor to Mr. Ευχαριστώ, κύριος Γκέρκε. Σας ευχαριστώ. Τώρα το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, θέλουμε να συνεχίσει να υφίσταται ως ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης. Πιστεύω ότι ο στόχος είναι φιλόδοξος γιατί πραγματικά έχει πολλούς ε, ευγενείς ε, στόχους αλλά για να υπάρξει μια στρατηγική αλλαγή θα πρέπει μια νέα περιοχή να ε, ξαναπλάσει τον εαυτό της και αυτό δεν μπορεί να γίνει από ψηλά. Θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους με αυτές τις γραφειοκρατικέ αναδιαρθρώσει τα χρήματα. Θα πρέπει να μείνουν στι περιοχέ, στα κράτη, στις περιφέρειες, στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μου επιμένει ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ επικουρικότητα, μεγαλύτερη ελευθερία για τα κράτη-μέλη και για τι περιφέρειε και λιγότερη γραφειοκρατία και στα πλαίσια τη γραφειοκρατική παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Χάρκιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την συγγήτρια. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμά έχουν τον ίδιο στόχο εδώ. Και ενώ υπάρχουν διαφορέ στην προσέγγιση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίες επί των οποίων θα συμφωνούμε όλοι. Διαφωνώ με τον κύριο Γκέρι και πρέπει να πω το Ταμείο Προσαρμογής στην Κοσμιοποίηση έχει να κάνει με αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν υπάρχει γιατί είναι κάτι καλό να κάνει κανείς, αλλά υπάρχει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη αρμοδιότητα στο εμπόριο. Και επομένως, όταν κάποιες από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε απευθείας και μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα προσπαθούμε στη συνέχεια να αναλαμβάνουμε μέτρα μετριασμού. Και σε αυτό στενίστε το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Σε ό,τι αφορά τι συμβιβαστικέ που παρουσίασε ήδη η συγκήτρια, υπάρχουν κάποια ίσονο σημασία ζητήματα, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνάντηση με του Κιώδης. Βέβαια υπάρχουν κάποια κύρια ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω συντομία. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία των ε, εκτοπισμένων θέσεων εργασία. Ε, συνολικά το παλιό ταμείο κάλυπτε 500 απολύσει, ε, το σημερινό είναι από 250 και πάνω, που είναι λογικό. Κάποιες από τις τροπολογίες πάνε κάτω από αυτό και αναζητούμε συμβιβασμούς μεταξύ 150 και 200. Η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ χαμηλός αυτός ο ρυθμός και θα σας πω γιατί. Γιατί πρέπει να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του ταμείου. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρές αγορές εργασίας. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να έχεις το 250 ως ελάχιστο. Ε, στο 50% των αιτήσεων μπορεί να έχουμε λιγότερους. Και στην ομάδα εργασία για το Ταμείο έχουμε δει πάρα πολλέ ε, αιτήσει ε, επιτυχημένε για κάτω από 250 πολυμένους. Έτσι λοιπόν το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε πρόσθεση των αριθμών στον ίδιο τομέα για να φτάσουμε τους 250. Είδαμε πριν τους χαρητήσεις που έρχονται από κράτου email, πριν τους χάρη στις κατασκευές ε, ή στην κλωστοεφαντουργία εταιρείε ε, που μπορεί να είχαν απολύσει 5-10 άτομα προσθέθηκαν όλα αυτά τα νούμερα προκειμένου να φτάσουμε στο κατόφλι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε όλα αυτά όταν μιλάμε για νούμερα. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία σε αυτό το σημείο. Επίσης, το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν ότι θα πρέπει να είναι ο συντελεστή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ. Γιατί δεν θα πρέπει να έχουμε ένα αυθαίρετο νούμερο του 70% όπως προτείνεται εδώ ή οποιοδήποτε άλλο νούμερο. Πάρα πολλά θέλω να πω, αλλά μακρηγόρησα. Και νομίζω ότι η συνάντηση των σκιωδών είναι το κατάλληλο σημείο να τα συζητήσουμε αυτά, το κατάλληλο φόρουμ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια πάντως για την καλή δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Ο κύριος Μιενταλόπες δεν βλέπω να είναι εδώ και δεν τον αντικαθιστά κανείς. η Βάνα από τους Πρασίνους. Ούτε αυτή είναι εδώ. Ούτε έχει αντικαταστάτη. Στην ε, Λάουρα Τζέα, παρακαλώ. Από τη FTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μαρία Ρένα για την εργασία της και κυρίως επειδή συμφωνούμε με την προσέγγισή της σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Κοσμοποίηση. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ε, υλοποίηση του Ταμείου αυτό στο δυνατόν πιο συγκεκριμένη, που θα πρέπει να υποστηρίξει τι επιχειρήσει που βιώνουν τα αποτελέσματα τη κρίση και τη παγκοσμιοποίηση. Οι δικέ μα τροπολογίε επικεντρώνονται σε κάποιε θεμελιώδε πτυχέ και είμαι ικανοποιημένη που η συνάδελφο ε, Αρένα συμφωνεί με τις δικές μας ε, σκέψεις. Καταρχήν, θέλω να τονίσω τη σημασία του να συμπεριλαμβούμε τον τριτογενή τομέα, όπου ο αντίκτυπος ε, της κρίσης έρχεται καθυστερημένα σε σχέση με τον δευτερογενή τομέα και να προστατεύσουμε αυτούς τους εργαζομένους καθώς και τους ε, ελεύθερους επαγγελματίες να σκεφτούμε να ε, καλύψουμε και τις επιχειρήσεις του τριτογενούς ε, τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και να έχουν την ε, δυνατότητα να ζητήσουν προληπτικά ε, κάποια δέσμευση πόρους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Ταμείο Προσαρμογής που Κοσμοποίηση να καλύπτει όλους τους εργαζομένους που έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου και είτε είναι εργαζόμενοι στον, ε, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή προσωρινοί εργαζόμενοι. Πρέπει να καλύψουμε όλες τις κατηγορίες. Είναι σημαντικό επίσης να μειώσουμε τους χρόνους αξιολόγησης ε, της αίτηση 40 ε, μέρες σε σχέση με τις 60 που προτείνονται από την Κομπισιόν. Κατά την άποψή μας για το κίνημα Τσινκουεστέλε είναι πιο σωστό ως χρονοδιάγραμμα. Επίσης, θα πρέπει να εργοποιήσουμε ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων, το οποίο θα εγγυάται μια έγκαιρη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν πιο πλήρη και ερμονισμένα στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά. Επικεντρωνόμαστε σήμερα σε αυτά τα στοιχεία που είναι τα πιο σημαντικά και είμαι σίγουρη ότι η δουλειά που θα κάνουμε μαζί με την εισηγήτρια που την ε, ευχαριστώ και για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην ανταλλαγή απόψεων για το ποιος έχει χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Ε, θα κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπισότο. Ο κύριος Μπισότο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να συγχωρήσετε την κυρία Μπισότο για την απουσία της. Ποιος θα μιλήσει όμως για τη δική σας ομάδα. Δεν είναι εδώ σκιώδη σας. Εντάξει. Να συνοψίσω λοιπόν λέγοντας ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Επασχόλησης θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη. Α, συγγνώμη. Η συγγήτρια θέλει να πει κάτι. Καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα. Σε σχέση με όσο υπόθηκαν και που είναι σημαντικά. Το πρώτο, σε σχέση με το υπόθηκαν από την κυρία Τούμ. σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τίτλος του Ταμείου, καθώς όμως το πεδίο της παρέμβασης δεν σχετίζεται μόνο με φαινόμενα παγκοσμιοποίησης, αλλά και με φαινόμενα μετάβασης, είτε μιλάμε για ενεργειακή ή τεχνολογική μετάβαση. Θεωρώ ότι να προσαρμόσουμε τον τίτλο στην πραγματικότητα του ταμείου που θα καλύπτει κάθε μετάβαση και όχι μόνο τη μετάβαση στην αποκοσμιοποίηση είναι κάτι κατάλληλο. Όπως είπα δεν είναι ε, ουσιαστικό, αλλά να έχουμε ένα ταμείο το οποίο έχει ε, τον τίτλο ε, τον κατάλληλο είναι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη ανησυχία που ακούστηκε από το ΕΛΚ, είναι σημαντικό να είναι πιο προσβάσιμο αυτό το ταμείο. Ναι, και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος της τροποποίησης που έχει θέσει η Κομισιόν ως προς το κατόφλι σε σχέση δηλαδή με τον αριθμό των απολυμμένων εργαζομένων, αλλά και σε ό,τι αφορά την περίοδο ε, που θα επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση στο Ταμείο. Θα προσθέσουμε και κάποιες τροπολογίες. Έχουμε αναφέρει τη δυνατότητα να ενημερώνεται περισσότερο τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις ικανότητες παρέμβασης. Πιστεύω ότι το θέμα της χρηματοδότησης, του ποσοστού της παρέμβασης είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ συμφωνώ να έχουμε μία ε, παραπομπή στο ECF συν, όμως πάντοτε συζητάτε το ποσοστό παρέμβασης ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ ε, και μπορούμε να έχουμε το χάρη 70% παρέμβασης, όμως δεν είναι παραδοσιακό αυτό το ταμείο, αλλά είναι ένα ταμείο αντίδρασης σε σχέση με τις απολύσεις όταν έχουμε μια επιχείρηση σαν αναδιάρθρωση. Σίγουρα θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, όπως είπε και η κυρία Χαρκίνη, σε ό,τι αφορά τα κατόφλια των εργαζομένων. Εμείς ε, εργαστήκαμε στο κατόφλι, επί του κατοφλίου το 250. Ε, δεν ε, υπάρχει τροπολογία για τη μείωση του κατοφλίου. Βέβαια, καθένας θα παρουσιάσει τις δικές του, τα δικά του επιχειρήματα και θα βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει φετιχισμός για το κατόφλι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου την πραγματικότητα επιτόπου, αλλά και την πραγματικότητα τη διοικητική, της διαχείρισης. Αν είναι πολύ χαμηλό το κατόφλι θα έχουμε δυσκολίες διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Χάρκιντζα, όταν απάντησε στον κύριο Γκέρικε, ότι τελικά ε, δεν είναι υπόθεση τη Ευρώπη. Μα ναι, είναι υπόθεση τη Ευρώπη, γιατί η μετάβαση είναι υπόθεση τη Ευρώπη. Αν έχουμε τεχνολογική, περιβαλλοντική μετάβαση, μετάβαση στην παγκοσμιοποίηση. Φυσικά η Ευρώπη εντάσσεται σε όλο αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα, ή συνέπειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητούν αλληλεγγύη και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι η αλληλεγγύη σε κάποιες περιοχές, σε κάποιους εργαζομένους που βιώνουν σήμερα δυσκολίες. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Και τέλος, κανένας δεν το ανέφερε, όμως στο πλαίσιο της ε, πρότασής μου έχω προτείνει να διευρύνουμε δηλαδή στο πλαίσιο της αντίδρασης, όχι στο πλαίσιο της πρόληψης, αλλά όταν κλείνει ε, μία ε, επιχείρηση ε, έχουν τραυματιστεί οι εργαζόμενοι επειδή έχουν χάσει και τη δουλειά τους συλλογικά αλλά και κάποιες περιοχές τραυματίζονται από, την δραστική, από το δραστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων και νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε ε, τους, ε, τις επιχειρήσεις ε, να συνεργαστούν. Στην Πορτογαλία είχαμε τον τομέα της κλωτοϊφαντουργίας όπου εργάζονται γυναίκες εκεί πάνω από 80%. Εγώ σέβομαι την πορτογαλική κυβέρνηση που έκανε την πρόταση αυτή να ε, εργαστούν οι γυναίκες σε παραδοσιακούς κλάδους για τις γυναίκες όπως παίρνουμε το σχάρι, τη φύλαξη των μικρών παιδιών, παιδιών, εκεί-εκεί βοηθή δεν θα ήταν σκόπιμο να εργαστούμε με, τις, ε, με τους τοπικούς φορείς της Βόρειας Πορτογαλίας για τις οικονομικές ευκαιρίες αυτής της περιοχής, ε, προκειμένου οι γυναίκες που έχουν τεχνογνωσία στην κλωστοεφαντουργία να μπορούν να εργαστούν σε άλλες βιομηχανίες παρά να τις τρέψουμε προς δημόσια απασχόληση. Ενώ θα υπήρχε δυνατότητα για ιδιωτική απασχόληση που να μην είναι ε, παραδοσιακά ε, επαγγέλματα γυναικεία, όπω λέγονται. Και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα στερεότυπα και στον Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Γιατί αν ε, εξισώνουμε, παραδείγματο χάρη, τη γυναίκα με τη φύλαξη των παιδιών και τον άντρα με την αεροαυπηγική, όχι. Θα πρέπει, ε, παραδείγματο χάρη, και οι γυναίκε που ασχολούνται στην κλωστή να μπορούν να απασχοληθούν στην Γιατί όχι και οι οικονομικοί φορείς ε, θα πρέπει να μάθουν από αυτά τα τραύματα, να συνεργαστούν και να βρουν τις καλύτερες ευκαιρίες ε, και να μην ακολουθούν την εύκολη οδό, να λένε ότι ο δημόσιος τομέας θα ε, απορροφήσει τις θέσεις απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα που κάποια στιγμή χάθηκαν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε το Ταμείο με ένα πολύ πιο δυναμικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν όχι δυναμικά από την πλευρά της Κομισιόν ε, ή από τη σκοπιά των εργαζομένων, αλλά με ένα πιο δυναμικό τρόπο ε, σε ό,τι αφορά ε, ουσιαστικά τις ικανότητες των περιοχών αυτή τη στιγμή. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει μια καλύτερη οικονομική ανάκαμψη των διάφορων ευρωπαϊκών περιφερειών σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αγένα. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 11. Α, ναι. Πριν περάσουμε στο σημείο 11, να πω ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Επασχόλησης στις 11 Νοεμβρίου για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στην παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, σημείο 11. Αποστασία των εργαζομένων από του κινδύνου που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνου ή μεταλλεξιογόνου παράγοντε κατά την εργασία. Ο λόγο στην κυρία Αγγέα, την κυρία Συγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν την ε, πρόταση οδηγία ε, την προστασία των εργαζομένων τη κοινή που συνδέεται με την έκθεση καρκινογόνου με τελεξιγόνου παράγοντε. Έφτασαν ε, από του σκιώδε ή από άλλε πολιτικέ ομάδε και εργάζομαι ήδη προκειμένου να μπορέσω να σα παρουσιάσω το συντομότερο μια συμβιβαστική πρόταση επί τη οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και εγώ κατέθεσα κάποιες, παρουσίασα κάποιες τροπολογίες Νομίζω στο σημείο που ίσως είναι το πιο πολύπλοκο της πρόσθεσης που αφορά τα κυταροστατικά φάρμακα. Υπήρξε ευρεία ανταλλαγή ε, email και υπήρξαν και πολλές συναντήσεις ε, και σε επίπεδο προσωπικού για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο. Και με πολύ ικανοποίηση μπορώ να πω ότι είμαστε κοντά στο να βρούμε ένα είδος συμβιβασμού που θα δεσμεύει την Κομισιόν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσει το παράρτημα 1 της οδηγίας με ένα κατάλογο επικίνδυνων φαρμάκων και των κυταροστατικών που είναι καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα και αυτό βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία αλλά και στις διαβουλεύσεις που είχαμε με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Ήταν σίγουρα ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σημείο, αλλά πιστεύω ότι με την καλή θέληση όλων θα μπορούσαμε και σε αυτό το θέμα να βρούμε μια συμφωνία και να μπορέσουμε και αυτές τις ουσίες να τις εντάξουμε ε, στην οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις και τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Και εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια κατάλληλη διατύπωση, ευθυγραμμιζόμενη και με ε, τις σκέψεις ε, σε δύο προηγούμενες ε, νομοθεσίες. Οι ειδικέ ε, ουσίες που έχουν ενταχθεί στην οδηγία, σημείωσα ότι ουσιαστικά έχουμε ισορροπία μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων και επομένως ε, είμαστε αρκετά κοντά στους, ε, στις οριακές τιμές που προτείνονται από την Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε επικοδομητική συζήτηση που να μας οδηγήσει σε έναν κατάλληλο συμβιβασμό. Θα στο κάδμιο και στο βυρίλιο βάσει των ε, όσων είδα από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν είναι οι μόνες ουσίες που τροποποιήθηκαν από κάποιους ε, εισηγητές, από κάποιους βουλευτές και επομένως απομακρύνονται κάπως από τα κατόφλια που προτείνονται από την Κομισιόν. Είδα ότι παρουσιάστηκαν και τροπολογίες ε, για τις εκπομπές αερίου δίζελ που είχαν παρουσιαστεί στο προηγούμενο μπάτς, δηλαδή στο δεύτερο μπάτς της οδηγίας και προληπτικά. Τώρα, θα χρειαζόταν να φτάσουμε ε, σε συμφωνία στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά θα παρουσιάσω τη θέση μας ε, για το σημείο αυτό, όμως το τρίτο μπάτς που θα προταθεί. Σίγουρα το δικό μου προσωπικό και το γραφείο μου είναι στη διάθεση όλων σας. Ζητώ μια προσπάθεια συνεργασίας περαιτέρω για να μπορέσουμε και σε αυτό το σημείο, το τμήμα της οδηγίας, να έχουμε το στο δυνατό αποτέλεσμα για να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων και να εγγυηθούμε βιώσιμα μέτρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μέγιστη δυνατή προστασία για τους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ. Thank you. Then I'll give the... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γολάν που είναι σκιώδης ηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εφόσον να δούμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδοχή ενωτήτων, batch. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό προσπαθεί να βρισκόμαστε σε μια συνεχή αναθεώρηση του ζητήματος. Βρισκόμαστε στο τρίτο μπάτ ε, τώρα. Θα υπάρχουν λιγότερε τροπολογίε, βέβαια, αν δεχτούμε τι τροπολογίε για τον ντίζελ. Αλλά είπε και η συγγήτρια ότι ε, θα μπορέσουμε να τις αποσύρουμε με μια συμφωνία για το δεύτερο μπάτς. Επομένω, ε, έχει γίνει σημαντική δουλειά από την εισηγήτρια για τις διάφορες τροπολογίες. Όπως είπατε, οι κατατοξικές ουσίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ε, άκουσα τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Εγώ από πλευρά μου ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τους εργαζομένους ε, από αυτές τις ουσίες, γιατί πολύ μεγάλος αριθμός ε, εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο καρκίνου, προσβολή τον καρκίνο λόγω της έκθεσης αυτές τις ε, ουσίες. Ε, αυτό προκύπτει ε, και από επιστημονικές μελέτες και από τους κοινωνικούς εταίρους. Ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο και τις οριακές τιμές, πρέπει να δούμε τι ισχύει και στις συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων, ιδίως σε περίπτωση που ευθυγραμμίζονται με επιστημονικές νομοδοτήσεις. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι η καταξιδότηση πράξης. Φοβάμαι ότι σε αυτό το σημείο μπορεί να ανοίξει κάπως ε, το κουτί της Πανδώρας. Γιατί οι καταξιδότητες πράξεις ε, υποτίθεται ότι πρέπει να τροποποιούν και να προσαρμόζουν μόνο μη ουσιώδη στοιχεία. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ουσιαστικά στοιχεία, όπως είναι οι τιμές αυτές, τα όρια που θα θέσουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, όλα αυτά να δερυθμίζονται με καταξιδότηση πράξης. Υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή, θα τα δούμε. Νομίζω ότι όπως και να έχει και με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις ε, έχουμε ήδη προετοιμαστεί και προθερμανθεί και μπορούμε τώρα να εργαστούμε ε, για να βρούμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε καλύτερα τους εργαζομένους. Thank you, Mr. Roland. I Ευχαριστούμε κύριε Γολά. Να πω κι εγώ δύο λόγια ως σκιώδης σε αυτή την έκθεση. Αρχικά να ευχαριστήσω την κυρία την κυρία Τζέα ε, και τους υπόλοιπους κοιόδης ε, για τα όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Για τις δικές μου τροπολογίες τώρα, μερικά σχόλια και ερωτήσεις. Πρώτον, έχω υποβάλει εκ νέου τις τροπολογίες μου για το CMD2, για τις ωρικές τιμές ε, για το diesel. Ελπίζω να μην χρειαστεί να εξετάσουμε αυτό το σημείο, γιατί ελπίζω να λυθεί αυτό το ζήτημα στην, ε, στον τριμερή διάλογο για το CMD2 αυτή την εβδομάδα. Αλλά πρέπει να υπάρξει μία οριακή τιμή για τις ε, εκπομπές diesel, γιατί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε αυτή την ουσία. Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος. Για τις κατροτοξικές ουσίες έχω υποβάλει τροπολογίε, ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ποιε ουσίε θα πρέπει να ενταχθούν στην οδηγία για τι καρκινογόνε και μεταξιογόνε ουσίε. Η κυρία Αντζέα είπε ότι πρόκειται για ένα νέο πεδίο. Πράγματι, είναι σοβαρό ζήτημα για του ε, εργαζομένου στον τομέα τη υγειονομική περίθαλψη και θέλω να διασφαλίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια. Φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους και να μην περιορίσουμε την πρόσβαση σε πολύ σημαντικά φάρμακα. Πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη. Έτσι, όπως και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ έχω επισημάνει ότι σε ό,τι αφορά τη φορμαλδεϊδή, η ιατρική χρήση της φορμαλίνης δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Αυτά προς διευκρίνηση, κατά κύριο λόγο. Βλέπω ότι και άλλοι συνάδελφοι συμφωνούν και ίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση. Τώρα, για το κάδμιο. Συχνά το συζητούμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί τις επαστομονικές νομοδοτήσεις. Δεν ε, βλέπω γιατί να τις απορρίψουμε. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε ε, υιοθετήσει. Σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν να τα υιοθετήσει και μάλιστα γρήγορα και η βιοπαρακολούθηση έχει προβληθεί ως σημαντικό πρότυπο ε, για την προστασία εργαζομένων. Κάποιοι μάλιστα ήρθαν σε επαφή μαζί μου και είπαν ότι θέλουν ε, να συνεχιστεί το biomonitoring και για αυτό το ζήτημα έχω κάποια ερωτήματα κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, ποιος θα είναι ο ρόλος της βιοπαρακολούθησης για το κάδμιο, της βιολογικής παρακολούθησης λοιπόν των ανθρώπων, ό,τι φορά το κάδμιο, αν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και πώς βλέπετε τη σύνδεση μεταξύ, ε, ε, του ορίου και τη συμπερίληψη τη βιολογική παρακολούθηση στην οδηγία. Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί να μην μπορούμε να συνδυάσουμε ε, την χαμηλή οριακή τιμή με την βιολογική παρακολούθηση. Εφόμενος αφόσον μάλλον η χαμηλή οριακή τιμή ε, επιβάλλει μια αλλαγή στην πράξη, ενώ η βιολογική παρακολούθηση εξετάζει τον αντίκτυπο. Γιατί λοιπόν η βιολογική παρακολούθηση να μην ε, εντάσσεται στην ε, εποπτεία της υγείας. Ελπίζω λοιπόν να ενταχθεί στις βέλτιστες πρακτικές αυτής της οδηγίας. Γι' αυτό θέλω να κατανοήσω καλύτερα κάποια πράγματα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει στοιχεία και σε αυτή την συνεδρίαση, αλλά και γραπτός, γιατί κάποιοι από εμά πρέπει να αποχωρήσουν ε, πριν το τέλος ε, της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Μάκιντάερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι έχουν παγιωθεί οι επιμέρους προσεγγίσεις και αυτό μας βοηθάει στη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος της έκθεσης στα χαμηλότερα δυνατά ε, επίπεδα, όμως είναι σημαντικό. Οι οριακές τιμές που θα θεσπίσουμε να είναι με, πρακτικά μετρήσιμες στον χώρο εργασίας. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά θέλω να το τονίσω και πάλι, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. επομένως τα επίπεδα, οι οριακές τιμές θα πρέπει να είναι μετρήσιμες εκεί όπου εργάζονται και πάντα θέλουμε να πετύχουμε τα, χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Επομένω, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ενεργά να επενδύουν ε, στην επιστήμη και να ενθαρρύνουμε ε, τις επιχειρήσεις να ε, προσπαθούν να πετύχουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Αλλά να μην θέτουμε αυθαίρετα επίπεδα, αυθαίρετες τιμές που δεν μπορούν να τηρηθούν βασική αρχή για του ε, συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ είναι ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση τροποποίηση των ωριακών τιμών θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια αυστηρή ε, διαδικασία ελέγχου ε, που ακολουθήθηκε και στην αρχή για τη θέσπιση των ορίων. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε, οποιασδήποτε επιπρόσθετες ουσίες θέλουμε ενδεχομένω να προσθέσουμε. Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε δύο ουσίες πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, για το βυρίλιο. Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι ε, το μεταβατικό URL, το 0,006 mg ανά τετραγωνικό μέτρο, προστατεύει την υγεία των εργαζομένων. Και από τεχνικής και οικονομικής άποψης ε, μπορεί να επιτευχθεί ε, στους περισσότερους κλάδους. Πριν από το τέλος της μεταδικής περίοδου υπήρξαν εκκλήσεις για μια υποχρεωτική δημόσια επισκόπηση σε ό,τι αφορά την ε, πρακτική εφαρμογή αυτών των ωριακών τιμών. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σαν ενδεχόμενο. Μετά, για την φορμαλδεΐδη. Να σας πω δύο πράγματα. Το ανέφερε και η Πρόεδρος προηγουμένως. Την φορμαλίνη έχω καταθέσει μια τροπολογία, νομίζω ότι είναι παριθμόν 69. Η φορμαλίνη αυτή είναι 37%, ένα διάλειμμα μάλλον 37% φορμαλδεΐδη ε, με νερό ως διαλύτη και χρησιμοποιείται γενικά για την ε, διατήρηση ανθρώπινων ιστών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τη ουσία αυτή στη διάγνωση νόσων. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα, ούτω ώστε η φορμαλίνη να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι γενικά θα όλοι μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Μετά, για την φορμαλίνη για τη χώρα μου είναι κάτι πολύ σημαντικό, μάλλον όχι για, για πολλές άλλες. Και αυτό γιατί στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά σύνηθες οι ε, συγγενείς του αποθανόντος να βλέπουν ε, ε, τη σωρό και μάλιστα αρκετά συχνά περνάνε δύο-τρεις εβδομάδες μέχρι την ταφή του νεκρού. Ξέρω ότι είναι ασυνήθιστο για άλλες χώρες, ιδίως στη Μεσόγειο, όπου η ταφή γίνεται πολύ γρήγορα. Αυτό δεν ισχύει στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πρέπει ε, να υπάρξουν απαραίτητες διαδικασίες ε, στη σωρό. Είναι λοιπόν σημαντική η μείωση ε, Τη έκθεση στη Φορμαδεϊδη. Γι' αυτό ε, και ο κλάδος εξετάζει πιθανά υποκατάστατα ή μείωση της χρήση φορμαλδεΐδης ε, στα προϊόντα ρήχευση και το έχουν ε, κατεβάσει το 0,5 αλλά δεν μπορούν να το κατεβάσουν το 0,3 αυτή τη στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να το λάβουμε υπόψη εάν τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι ασφαλές. Επομένω, η ε, μελέτη αντικτύπου για την αρχική πρόταση σε ό,τι αφορά τη φορμαλδέιδη επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην χρήση της φορμαλδεΐδης, στις κόλλες και στην συντήρηση ξύλου. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ε, ταρίχευση ε, δεν έχει καλυφθεί αυτό το ζήτημα επαρκώς. Γι' αυτό θα ήθελα η συγγήτρια και οι ε, να εξετάσουν ενδεχόμενο μεταβατικής περίοδου για αυτή την πολύ συγκεκριμένη χρήση της φορμαλδέιδης. Σίγουρα θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς στη συνεδρίαση των σκιωδών. Και φυσικά θα υπάρξει αγαστή συνεργασία όπως πάντα. Ωραία. Ο κύριος Καλβέ Σαμπον έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που είναι πολύ επικοδομητικά. Γιατί ποιος δεν θα συμφωνήσει με το να βελτιώσουμε την υγεία των εργαζομένων, δηλαδή την υγεία όλων ημών κατά κάποιο τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο μας επιτρέπουν οι τεχνικοί και, οι... και τα οικονομικά. Και εγώ νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό του αποκαλούμενου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτή την οδηγία και δεσμευόμαστε στο να τη διαπραγματευτούμε για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα για τους εργαζομένους Πιστεύουμε ότι το έργο της εισηγήτριας είναι εξαιρετικό. Θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση εργασίας. Επίσης, συνάδει με όσα έχουν υλοποιηθεί και είναι πολύ καλό να υπάρχει μια συνέχεια με το batch 2 του κυρίου Ρολάν. Και αυτό οδηγεί, περίπτωση χάρη, στο συνέχιση του έργου αυτού του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα του ντίζελ που συνεχίζει να υποστηρίζει η δική μου ομάδα ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη έχει να κάνει με τις ευαισθησίες του τριμερούς διαλόγου για τον ΠΑΤΣ 2. Και φυσικά χωρίς να ξεχνάμε τα θέματα που μπορεί να ξανατεθούν στις συζητήσεις για τον ΠΑΤΣ 3. Πάντοτε το λέγαμε ότι είναι σημαντικό για μας, γιατί πρέπει να είμαστε σοβαροί, ότι τα όρια θα πρέπει να τίθεται βάσει μιας διαδικασίας ε, που θα βασίζεται στα επιστημονικά στοιχεία και στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. θα πρέπει αυτά να είναι αξιόπιστα τη στιγμή που θα εφαρμοστούν και σε τεχνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, η επιστήμη συνεχώς εξελίσσεται και επιτρέπει κάθε φορά να ενιχνεύουμε περισσότερα. Εγώ όταν ήμουν διευθυντής ε, ανάπτυξης σε ένα ορυχείο ε, ουσιαστικά δεν ε, είχε να κάνει με το τι ε, έβγαινε στην ατμόσφαιρα. Το θέμα ήταν ε, τι μπορούσαμε να μετρήσουμε. Σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε 100 φορές περισσότερο με τις νέες συσκευέ. Εργαζόμουν σε ορχή για Όμως ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το θέμα των εργαζομένων, των θέσεων εργασίας. Και ξέρετε, το βέλτιστο πολλές φορές μπορεί να είναι εχθρός του καλού. Επομένως, μια ισορροπημένη κατάσταση θα είναι να έχουμε και χρόνο για την προσαρμογή. Και επίσης ε, να μπορούμε και από οικονομική σκοπιά να αντέχουμε αυτό το ρυθμό. Και όσα λέει η κυρία Τζέα, νομίζω δεν αντιτίθεται σε αυτές τις ιδέες, γιατί τελικά η έκθεση των ατόμων θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις σε υλικά που δεν επιτρέπουν την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Σίγουρα στις τροπολογίες μας εμείς θα έχουμε και κατά νου τον αντίκτυπο στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Η συγκήτρια, πέρα από το θέμα του ντίζελ που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, προσθέτει και ζητά να ληφθούν υπόψη τα κυτάροτοξικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τους εργαζομένους που χειρίζονται τα φάρμακα για τις ογκολογικές θεραπείες. Ούτε μπορούν να γίνουν μάρτυρες οι άνθρωποι αυτοί, ούτε μπορούμε να έχουμε παρενέργειες γιατί μπορεί τελικά να έχουμε λιγότερου εργαζομένου στον τομέα επειδή θα φοβούνται. Όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την υγεία όλη τη κοινωνία. Επομένω, στι τροπολογίε μου, λέγοντα ότι μου φαίνεται καλή η ιδέα τη κυρία Ατζέα, θα τονίσω τις ε, διαφορές που υπάρχουν σύμφωνα με τους επιστήμονες μεταξύ διάφορων κυταροτοξικών και της ε, επιστημονικά ορθής θεμελίωσης όσων είναι επικίνδυνων. Δηλαδή τα επίπεδα που έχουμε σε κάθε κυταρτοξικό φάρμακο. Δεν θέλουμε τώρα πραγματικά να κρούσουμε τον κοντά του κινδύνου και να αρχίσουν ξαφνικά να φοβούνται οι εργαζόμενοι. θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Έτσι λοιπόν, εντός αυτής της επικοδομητικής γραμμής και βάσει της εξαιρετικής δουλειάς της κυρίας Ατζέα, εγώ νομίζω ότι θα κινηθούν δικέ μου τροπολογίε και τροπολογίε του Άλντε και ότι τελικά θα έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο για να διαπραγματευτούμε στους τριμερεί διαλόγου. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ. Κυρία Λάμπερτ για του ε, πρασίνου. Okay, thank you. I'm speaking. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στον με του ε, του συναδέλφου που λείπει κάποια βασικά στοιχεία. Ένα από τα βασικά στοιχεία για μας λοιπόν είναι οι ουσίες που κατηγοριοποιούνται ε, στις καρκινογόνες μεταξυγόνες ουσίες ε, βάσει του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού. Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη αξιολόγηση κινδύνου σε αφορά την έκθεση σε συντελεστή πάνω από 1 προς 2.500. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν και μια ρήτρα αναθεώρηση στην πρόταση για την ομάδα μας. Η βιολογική παρακολούθηση που προτείνει η συγγήτρια μας βρίσκει αντίθετους. Θα θέλαμε επίσης πιο σύντομες ε, μεταβατικές περιόδους που να συνάδουν με το γενικότερο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί ήδη από τους κοινωνικού εταίρους. Και για ορισμένα από τα άλλα ζητήματα, φυσικά θα τα μεταφέρουμε στη συνάδελφο Καρή Μαντέλη για να τα λάβει υπόψη. Αυτά από μας. Ευχαριστώ. Merci. Ε, pour e NF, Madame Melin. Oui. Κύριε Μελάν από το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και Ω εισηγήτρια από την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα εξετάσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να σας πω ότι ε, για πρώτη φορά θεωρώ ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο, γιατί μετά από τι ε, μακρέ συζητήσει που κάναμε στου δύο πρώτου ε, γύρου σε ό,τι αφορά τις καρκινογόνε ουσίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη την ε, συσσωροπία των συμφερόντων των εργαζομένων, αλλά και τα συμφέροντα των εργοδοτών, οι οποίοι σε κάποιε περιπτώσει δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τι προδιαγραφέ και να επανεπενδύσουν. Θα θέλαμε λοιπόν να κοιτάξουμε και πιο στενά, πιο αντελεχώ τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία χορήγησαν οι 27 χώρε μέλη για τι 7 ουσίες τη οδηγία. Ήταν τόσο κοντινά που δεν είχε νόημα να πάμε παραπάνω σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν καλές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Ενδεχομένω ε, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Σε ό,τι αφορά, και θα ξέρετε, μια και συμμετείχατε στην ψηφοφορία, υπήρχαν ε, κάποιες προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν με τρόπο αντιδημοκρατικό σε ό,τι αφορά το φάκελο αυτό που καταρτίστηκε ουσιαστικά από τροπολογίε των διαφορών ομάδων. Κρίμα γιατί η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή Περιβάλλοντο για τρίτη φορά δεν έδωσε την απάντηση που θα έπρεπε να δώσει στην Επιτροπή Απασχόληση. Γιατί αν κάποιε ουσίε έρθουν σε επαφή με το δέρμα, φλωρανελίνη και φλωρμαλδεΐδη, ο περιβαλλοντικός παράγοντας ε, παραμένει σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο βερίλιο όμως ε, και στο κάδμιο που απαντώται στην ατμόσφαιρα ακόμα και 20-30 χρόνια μετά τη χρήση τους σε μεταλλουργικές εταιρείε, ε, σε κατασκευαστικές. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζουμε την εξή δυσκολία ο εργαζόμενος όταν ε, ζητά να αναγνωριστεί η επαγγελματική του ασθένεια, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ του περιβαλλοντικού παράγοντα, της ασθένειάς τους, της πάθησής του και της εργασίας τους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επικριθούμε στις ουσίες όπου δεν υπάρχει μεγάλη συζήτηση ως προς τον καρκινογόνο αντίκτυπο, ότι όπου γίνεται αποδεκτός αυτός ο αντίκτυπος, ότι η συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι κρίμα που κάθε φορά προσπαθούμε να τροποποιήσουμε, παρά το γεγονός ότι φυσικά πρέπει να το συζητήσουμε, την οδηγία αυτή με ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη χρήση τους και έχω υπόψη μου και διάφορες ουσίες φαρμακευτικές ε, σε ό,τι αφορά τις ουσίες εκείνες ε, οι οποίες έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο και το τοξικές κτλ. που αφορούν όλους τους ανθρώπους και μέσω των καυσαρίων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, ουσίες που μας προτείνονται και κοιτάξτε, Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τρέχουσα θετία. Να σας πω ότι τα όρια του καρκίνου και των παθήσεων δεν είναι πολιτικά και δεν θα πρέπει να μην ακούμε τους ε, συναδέλφους οι οποίοι όμως ενδεχομένω να έχουν και άλλα συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Και τα θέματα τα οποία έθιξε η πρόεδρος η κυρία Μουσκάτ θα υπάρξει απάντηση γραπτά αλλά αν θέλει να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει ήδη, μπορείτε. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλησπέρα. Κρίστεν Κάιντρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ε, έκθεση, για το σχέδιο έκθεση. Το διαβάσαμε με προσοχή και φυσικά χαιρόμαστε που δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγέ στις προτινόμενε οριακέ τιμέ. Φυσικά για την μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο στενά τα πράγματα και βασικά να σας πούμε ότι και εμεί διακρίνουμε το φω στην ακρίβεια του τούνελ σε ό,τι αφορά τον ντίζελ. Μακάρι λοιπόν να σημειωθεί πρόοδο εκεί. Φυσικά μας απασχολούν τα το τοξικά φάρμακα. Δεν ε, υποβάλαμε σχετική πρόταση για κάποιους λόγους. Δεν λάβαμε και δεν συμπεριλάβαμε τα επικίνδυνα φάρμακα εδώ, γιατί καταρχάς υπάρχει κατάλογος των ε, φάρμακων σε ό,τι αφορά τα καρκινογόνα, τα οποία ρυθμίζονται από ειδική διαδικασία. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστός και συνεκτικός κατάλογος των ε, ουσιών αυτών και δεν υπάρχει και επιστημονική ευρωπαϊκή ε, αξιολόγηση των φαρμάκων αυτών. Δεν υπάρχει μελέτη δεκτύπου σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό, οικονομικό αντίκτυπο. Και επίσης δεν είμαστε βέβαιοι ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πώς είναι η σωστή οδηγία αυτή για τα καρκινογόνα, γιατί υπάρχουν και άλλες οδηγίες οι οποίες ενδεχομένω να είναι πιο ανταδειγμένες. Θα πρέπει να ενημερώσουμε επίσης και τις κατευθυντήριες γραμμές. Και κοιτάξτε, έχοντας ολοκληρώσει την εργασία για το diesel τις τελευταίες ε, εβδομάδες, μήνες, σχεδόν ένα χρόνο μαζί σας, ανησυχώ, ανησυχώ ότι είναι λίγο πρόωρο να θέσουμε στο τραπέζι και στην τρίτη πρόταση τις ουσίες αυτές. Ο πρόεδρος Γιούγκερ στην επίστολη πρόθεση προς τον Σεμπάστιαν Αγκόσιν και στον Αντώνη Ταγιάννη ανέφερε ότι το, ο φάκελος αυτός, η τρίτη ενότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα θετία για τα τοξικά φάρμακα, αλλά προφανώς και τα παίρνουμε στα σοβαρά και μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Θα δούμε τι θα προκύψει και από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τα θέματα που ακούσαμε για το κάδμιο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μας έδωσε δύο ε, λύσεις, ε, επίπεδο 1 και επίπεδο 4, ανάλογα με την ε, βιοεποπτεία σε ό,τι αφορά και την οδηγία για τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα, γιατί η οδηγία αυτή δεν μπορεί να τα συμπεριλάβει. Γιατί η οδηγία αυτή έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα και αυτό που αναπνέει ο εργαζόμενος και την πρόσληψη μέσω του δέρματος μας συμβούλεψε λοιπόν η νομική υπηρεσία να μην συμπεριλάβουμε αυτές τις ουσίες στο κάτμιο. Και επίσης αυτή η πρόταση υποβλήθηκε και καθυστερημένα. Θα δούμε λοιπόν. Για το κάδμιο. Μας σύστησε λοιπόν η νομική υπηρεσία να μην συμπεριληφθεί στην βιοπαρακολούθηση στην ενότητα αυτή τη οδηγία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και την απόψη τη νομική υπηρεσία. Υπήρξαν και προτάσει από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την βιοπαρακολούθηση για να υπάρξει μεγαλύτερη ε, οριακή τιμή και να είναι λιγότερο αυστηρά λοιπόν τα πρότυπα. Αλλά όπως και να έχει, εμεί πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο στα κράτη-μέλη. Η συζήτηση για τη φορμαδεΐδη. Επίσης έγινε αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή συμβουλευτική και σε ό,τι αφορά και την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στον Εμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. έξω όσων ε, καταλάβαμε, θα δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρξει μια σωστή εξαίρεση ή πρόβλεψη απόκλησης και για το βαρέλιο και για άλλες ουσίες. Έγινε συζητήσεις επί μακρόν, έγιναν και κάποιες προτάσεις από πλευρά σα για να είναι λίγο πιο εκτενήσει ή λιγότερο εκτενήσει η λιγοτερο εκτενή η προταση Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική σα τοποθέτηση όταν και θα αποφασίσετε. Τα σημειώνουμε ωστόσο όλα αυτά και προφανώς και θα περάσετε μερή διάλογο. Η σημασία διενεργίας μελέτη αντικτύπου και της ε, σωστής επιστημονικής ε, αξιολόγησης. Ε, συμφωνώ απόλυτα για τα οξυτοξικά φάρμακα δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Έχουμε την πρόταση ΆΙΑΚ και τα συμπεράσματα για τα το, φάρμακα σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες τους, τις καρκινογόνες ιδιότητες τους. Αυτά λοιπόν τα σχόλιά μου στην παρούσα φάση και προσβλέπω στην μελλοντική εκδοχή της έκθεσης. Κάποιες άλλες ε, ερωτήσεις σας θα σας τις απαντήσω γραπτά αν σας πειράζει γιατί είναι πολύ τεχνικές και πρέπει να συμβουλευτώ τους συναδέλφους πρώτου τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει δουλειά. 20 Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία και μέχρι τότε θα γίνουν διάφορες συνεδριάσεις ε, σχεδόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το θέμα της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής λειτουργίας σταθεροποίησης επενδύσεων και να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Καλβέ Σομπον, που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις, η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται στο εξή πλαίσιο, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σημαντική έλλειψη επενδύσεων που αποδυναμώνουν σημαντικά την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ένωσης που αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ας θυμηθούμε ότι αυτό το γελίο πράγμα που ονομάζεται προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το 0,9% ίσως 1%, ούτε καν χρησιμοποιείται για ευρωπαϊκέ επενδύσει γιατί δεν μένουν χρήματα. Δηλαδή, όταν έχουμε αφαιρέσει τι δαπάνε λειτουργία και τη κοινή αγροτική πολιτική, τα κονδύλια είναι αλληλεγγύη, αλλά για εθνικά προγράμματα, όχι για επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν 25-35% μεσοπονδιακού προπολογισμού για κάτι τέτοιο από την άλλη. Έτσι λοιπόν το να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση είναι χαριτωμένο, έτσι. Η παγκόσμια κρίση μας έχει δείξει τους τεράστιους περιορισμούς των μέσων που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, ξεχωριστά, μεμονωμένα, που βασίζονται ουσιαστικά αποκλειστικά στην ε, ενιαία νομισματική πολιτική. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία σε καμία περίπτωση για να μετριάσει μεγάλους ασμέτρους κλειδονισμούς, ούτε για να εγγυηθεί αποτελεσματικά την διατήρηση των ε, επέδων των δημοσίων επενδύσεων στα κράτη-μέλη. Πέρα από τον εμβαθύνει και να παγιώσει, θα πρέπει να καταστήσει ε, να κατασταθεί συγγνώμη, ρεαλιστική οικονομική και νομισματική ένωση, χρειάζονται αποφασιστικές δράσεις, όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και την υποστήριξη δημοσιονομικών μέτρων και μέτρων συντονισμού της πολιτικής των πολιτικών της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων που προτείνεται πρέπει να βοηθήσει να σταθεροποιηθούν οι δημόσιες επενδύσεις με ε, μορφή επέσπαση των ε, συμφερόντων κρατών μελών ε, που ουσιαστικά πλήττονται από ασύμετρους κλειδονισμούς όταν δεν αρκούν τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκυρίες όταν δεν υπάρχει φυσικά εθνική νομισματική πολιτική και όταν ο συντονισμός των φορολογικών δημοσιονομικών πολιτικών έχουν φτάσει στα όρια τους και δεν γίνονται πλέον ανεκτές κοινωνικά. Εκεί θα πρέπει να παρεμβαίνει αυτό το Ταμείο Σταθεροποίησης Επενδύσεων. Η θέση του εισηγητή είναι ότι πάντοτε καλύτερο είναι να υπάρχει κάτι από το τίποτα. Και καθώς ε, οδεύει προ την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε φυσικά να το υποστηρίξουμε. Προφανώ εγώ θα προτείνω στην ομάδα να το υποστηρίξει. Βέβαια πρέπει να δηλώνουμε και τις ανεπάρκειες, δηλαδή να μην πιστεύετε ότι με αυτό έχουν λυθεί τα θεμελιώδη προβλήματα της Νομισματικής Ένωσης, αλλά τέλος πάντων καλύτερα να κάνουμε κάτι παρά τίποτα και μακροπρόθεσμα αυτό το σύστημα φυσικά θα βοηθούσε στο να έχουμε περισσότερη απασχόληση και να καταπολμηθούν και οι αντικυκλικές πολιτικές. Όμως εδώ έχουμε δύο προβλήματα τα οποία εγώ θα τονίσω. Δεν ξέρουμε τη βοήθεια όλων σας ίσως. Καταρχήν, το ποσό που προβλέπετε των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι σχεδόν το ίμιση, πάνω κάτω το ίμιση της διάσωσης μιας χώρας, όχι πολύ μεγάλης όπως η Ιρλανδία. Αν ε, γίνω πολύ επιθετικός θα έλεγα ότι είναι γελίο το ποσό αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ας προσπαθήσω να μην είμαι. Επιθετικός είναι ξεκάθαρα ανεπαρκές το ποσό αυτό και θα έπρεπε να μάθουμε και κάτι από τα νούμερα της πρόσφατης κρίσης. Και κατόπιν θα σας προτείνω να παρέμβουμε στα κριτήρια επιλογής. Είναι αυστηρά αυτά που εκτίθενται, γιατί ουσιαστικά την ε, ανεργία την αντιμετωπίσουν με κάποια κριτήρια που είναι επιστημονικά σωστά, ωραία, είναι θεμελιώδε στο θέμα της ανεργίας και πρέπει να δούμε πότε είναι διαθροτική ανεργία και φυσικά πότε χρειάζεται μία ενίσχυση στο κράτος στη σταθεροποίηση των επενδύσεων. Αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Έχουμε πάρα πολύ ευπαθή κατάσταση στην Νομισματική Ένωση και στην Ευρώπη και μία από αυτές είναι η ε, μεγάλη αύξηση των ενισοτήτων σε κάποιες χώρες και επίσης η απαράδεκτη αύξηση της φτώχειας και φυσικά αυτά συνδέονται. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να έχουμε τον εμπλουτισμό των κριτηρίων με πολύ ξεκάθαρα κοινωνικά κριτήρια γιατί είναι λάθος να σκεφτόμαστε ότι η ενίσχυση Ε, ουσιαστικά πρέπει να γίνεται μόνο σε οικονομικό επίπεδο ή ότι η Ένωση Οικονομική και Νομισματική είναι πρόβλημα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να υπάρχει νομισματική ένωση όταν δεν υπάρχει πολιτική ένωση. Όταν δεν υπάρχει πολιτική ένωση, η νομισματική ένωση χάθηκε. Έτσι λοιπόν αυτό τι σημαίνει ότι θα μας απασχολήσουν εδώ τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί είμαστε και Επιτροπή απασχόληση. Τη στιγμή που θα προωθήσουμε την πιο διευρυμένη χρήση και λειτουργικότητα του Ταμείου αυτού. Μου λέει ο πρόεδρος ότι έχω μακρηγορήσει πολύ και πρέπει να περιοριστώ. Τέλο πάντων, τα ουσιαστικά τα παρουσίασα. Διαβάστε παρακαλώ και τις δικές μου συνεισφορές, περιμένω και τις δικές σας και σίγουρα θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την έκθεσή μας. Η πρόθεση θα είναι να καταστεί το Ταμείο αυτό όσο το δυνατό πιο λειτουργικό ως προς την απασχόληση και ως προς την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Και θα σταματήσω εδώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Σκιώδης. Εξ ονόματος του Έλκεν, ο κύριος ε, Τιτιές Ροφουά δεν είναι εδώ. Στη συγγνώμη για την απουσία του, όμως μου μετέφερε την ανακοίνωσή του. Το ΕΛΚ θέλει να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός, αντίστοιχος με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης των Επενδύσεων, για την προστασία των επενδύσεων των κρατών μελών σε καιρούς κρίσης επιθυμεί μια Ευρώπη που ε, προστατεύει και ως εκ τούτου είναι ευνοϊκά διακείμενο ω προς την ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να θεσπίσει ένα τέτοιο μηχανισμό που θα μετριάσει τους ε, οικονομικούς κραδασμού. Ωστόσο, το προσχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει και αρκετά προβληματικά στοιχεία κατά τη γνώμη του που υπερβαίνουν την αρχική πρόταση. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο σημεία. ότι ε, κινητοποιούνται οι μηχανισμοί και σε περίπτωση μετριασμού, αλλά και σε άλλε περιπτώσει που αλλάζουν ε, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Δεύτερον, το ΕΛΚ ε, αντιτίθεται σε πιθανή αύξηση των κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το Ταμείο. Ο προπολογισμό θα πρέπει να έχει ως στόχο την στήριξη χρηματοδότηση των βασικών επενδυτικών προγραμμάτων που θα οδηγούν σε απαραίτητε διευθυντικέ μεταρρυθμίσει. Ε, για το ΕΛΚ, τα κονδύλια θα πρέπει να στηρίζουν στο βαθμό του δυνατού ε, προγράμματα κλειδιά που θα ε, τονώνουν την αγορά απασχόληση και θέλει διευκρινήσει σε ό,τι αφορά τον εισηγητή και αν στο μέλλον επιθυμεί μια θέσπιση μακροοικονομικού επενδυτικού μηχανισμού τι εννοεί δηλαδή ακριβώς ο εισηγητής με αυτή την ε, τοποθέτηση, γιατί ήδη αυτό είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης των Επενδύσεων και αφετέρου. Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος για περισσότερου μηχανισμού και περισσότερε επιλογέ στα κράτη-μέλη. Επομένω, ο Σκιώδη εισηγητή θα ήθελε να έχει περισσότερε διευκρινήσει σε ό,τι αφορά αυτό το στοιχείο. Pour de Didier euh, Geoffroy. Αυτά μου μετέφερε ο κύριο Διδιέ Ζοφχουά. Για τους σοσιαλιστές, οι Άγνε τώρα. Επίσης, εξ του σχεώδους εισηγητή που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, μου έδωσε τι σημειώσει του για την εν λόγω πρόταση. Βέβαια, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε των ε, ζητημάτων που άπτονται των αρμοδοτήτων τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η ομάδα μου έχει όμω κάποιε σκέψει για την απρόταση. Αρχικά, οι στόχοι αυτού του νέου ταμείου θα πρέπει να διευκρινιστούν και να οριστικοποιηθούν περαιτέρω σε σχέση και με τα άλλα θεσμικά όργανα που υπάρχουν. Η δημιουργία μια τέτοια λειτουργία σταθεροποίηση είναι πολύ καλή πρόταση για την καλύτερη αξιοποίηση του ενωσιακού προπολογισμού, για την αύξηση τη ανθεκτικότητα των αλληλεξαρτημένων οικονομιών μα και θα συμβάλλει και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Πολύ καλό λοιπόν αυτό, πολύ θετικό. Όμω η κοινωνική συνοχή δεν αφορά μόνο τον ε, συντελεστή απασχόληση, κατάρτιση. Ε, γι' αυτό θα θέλαμε ο στόχο, τον, τη συμπερίληψη με καλύτερο τρόπο του στόχου του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τα κριτήρια δημοσίων επενδύσεων. Και ως προς αυτό συμμεριζόμαστε τη γνώμη του εισηγητή. Δεύτερον, η αιρεσιμότητα που προκύπτει από τα κριτήρια επιλεξιμότητας θεωρούμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί και τα κράτη-μέλη που χρειάζονται περισσότερο την ε, σταθεροποίηση βλέπουμε ότι συνήθως ε, έχουν ενταχθεί σε ε, προγράμματα προσαρμογής ή διαδικασίες ανισοτήτων. Μετά, τα κριτήρια αξιοποιούν μόνο εθνικά στοιχεία απασχόλησης Πρέπει όμω να βάλει λάβουμε υπόψη και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα θα οδηγούσε στην ενεργοποίηση αυτών αυτού του μηχανισμού όταν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο. Να μην χρησιμοποιούνται δηλαδή μόνο τα εθνικά στοιχεία ενεργείας, αλλά και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Point ε, of reference. Ε, if this instrument intends to Εάν θέλουμε λοιπόν αυτός ο μηχανισμός να συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρος ανεργίας που θα καταδεικνύει αν θα υπάρξει περαιτέρω κοινωνική συνοχή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, μόνο ο συντελεστής ανεργίας θα πρέπει να αξιοποιείται για την αξιολόγηση ασύμετρων ε, κραδασμών. Μετά, ο μηχανισμό δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο καθεστώ προστασία επενδύσεων, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να υπάρχει και ένα καθεστώ επιδόματο ανεργία, όταν το ποσοστό ανεργίας ή μάλλον όταν θέλουμε να ε, στηρίξουμε ε, τα καθεστώτα επιδομάτων ενεργείας στα κράτη-μέλη. Τέλος, ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, διασφαλίζεται και στη διακυβέρνηση του μηχανισμού, ιδίως ό,τι αφορά την παρακολούθηση της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των δημοσίων επενδύσεων. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτό θα, το κάνει μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Ενώ εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να εμπλέκεται το Κοινοβούλιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον εισηγητή και θα συνεργαστούμε μαζί του για να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω η πρόταση. Euh, Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Καλβεσσαμπά. Αυτό το Ταμείο Σταθεροποίησης Επενδύσεων ουσιαστικά ε, έχει σκοπό να καταπολεμήσει ασύμμετρου συγκλονισμού στην ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση που έχουν αρνητικό αντικτύπο σε διάφορε περιφερειέ ή έχουν αρνητικό αντικτύπο και μεγαλύτερε συνέπειε για κάποια περιφέρεια, για κάποιο κράτο μέλο. Έτσι ήθιστα Δυστυχώ, ε, τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν ε, είναι τα κατάλληλα για να απορροφηθούν αυτοί οι κλειδονισμοί. Γιατί αντιπαραθέτουν ε, τις περιφέρειες και έχουν να κάνουν και με τις ίδιες τιμές στο ένα κράτος. Δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε έτσι τις αυτού αυτούς κλειδονισμούς. Δεν πρόκειται να αρκέσει αυτή η παράμετρος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω να απευθύνω αυτή την ερώτηση σε ό,τι αφορά τους συνηθισμένους επιστημονικούς όρους και ορισμούς. Ε, γιατί δεν χρησιμοποίησα τους ε, αναγνωρισμένους όρους και ορισμούς και έφτιαξα δικούς τη. ή μήπως είναι θέμα μετάφρασης. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά την ε, έλλειψη διαγωνιστικότητας της χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό οφείλεται στη μήτηρη των κριτηρίων του Μάστρεχτ. Αν λοιπόν τα κράτη που το πετυχαίνουν αυτό, πώς θα το λύσουμε, η σύγκληση μέσω μεταφοράς, τι θα συμβεί σε μία ύφεση, οι ισχυροί θα έχουν μείωση των επενδύσεων τους και η διαφορά θα την πληρώσουν τέτοια ταμεία. Η αρχή των δημόσιων επενδύσεων επίσης ορίζεται ο μέσος όρος είναι 3% σύμφωνα με τον ΑΣΑ. Μιλάμε για μεγάλα ποσά και σύμφωνα με τις ε, εκτιμήσεις αυτές ε, και ο Καλβέσιο ανέφερε την Ιταλία είναι 45 εκατομμύρια ευρώ και σε μια άλλη κρίση δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε υποστήριξη 30 εκατομμυρίων. Ο εισηγητής ε, φαίνεται ότι να γνωρίζει αυτό και το ανέφερε. το 2025 να υπάρξει αύξηση του ποσού, όχι μετά από ανεξάρτητη ε, με, μεταρρύθμιση, αλλά από μεταρρύθμιση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να εκτιμήσει τη δική της ε, ε, εργασία και μετά να δούμε τι θα προκύψει. Εδώ μας λείπει και θα πρέπει να συμφωνήσω με την συνάδελφο από τους Σοσιαλδημοκράτες, την κυρία Γιονγκέριους. Λείπει ο κοινοπλαστικός έλεγχος και πολύ αντιχειρωτώμε γιατί δεν απαιτούμε σωστό κοινοπλευτικό έλεγχο. Αυτό σίγουρα θεωρώ ότι μπορούμε να το συμπληρώσουμε μέσω τροπολογιών. Γιατί το ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο το οποίο θέλουμε να δημιουργηθεί μέσω διακυβερνητικών αποφάσεων. Να σκεφτούμε λοιπόν πού θα ενταχθεί αυτό ο κοινοβουλευτικό έλεγχο εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από τι Εθνικέ Βουλέ. Τώρα, η έκθεση εκτίμησης του τη Ευρωπαϊκή Λειτουργία Αγαπήση Επενδύσεων θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το δημοκρατικό έλεγχο και θα ήθελα να ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει και δεν προτείνει αλλαγή των συνθηκών για τη δημιουργία αυτού του ταμείου, γιατί το η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίηση Επενδύσεων θα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι στην άμεση αρμοδιότητά τη. Μήπω θα προκύψει ένας κυκαιώνας ευρωπαϊκών διακρατικών ε, συμφωνιών αυτό προφανώς ε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και στον Ευρωπαίο πολίτη. Πώς να το εξηγήσουμε αφού είναι τελείω αδιαφανέ. Ε, αυτό λοιπόν το Ταμείο ε, Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίηση Επενδύσεων θα καταλήξει να είναι ένα ακόμα αρκτικό λέξο. Κανείς Ευρωπαίος πολίτης δεν θα καταλαβαίνει ούτε το νομικό καθεστώ, ούτε τη λειτουργία τη λειτουργία του Ταμείου αυτού. Και θεωρώ ότι δημιουργούμε όλο και πιο πολλά και περίπλοκα οικοδομήματα και σύνθετα νομικά τέρατα τα οποία δεν τα κανένα. κανένας. Και άλλη μια ερώτηση να κάνω προς τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αγγλική μετάφραση. Αναφέρεται maximum amount of loans και ότι το υπόλοιπα, οι υπόλοιπε πιστώσεις που θα, χορηγούν, θα χορηγούνται προς τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα είναι 30 εκατομμύρια επί της αρχής. In principle, τι εννοείται με αυτό το in principle. Ίσως να γνωρίζετε κάποια ανέκδοτα που λένε ότι ναι, επί της αρχής ναι, αλλά θα ήθελα λοιπόν να τα απορρίψουμε αυτές τις προτάσεις και θα ήθελα να υποβάλει άλλα κριτήρια ενεργοποίησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή και ζητώ από όλους τους συναδέλφους μου να φροντίσουν να υπάρξει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αν θέλετε να ενισχύσετε την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό μέσω αλλαγή των συνθήκων. Θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε και παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξη ότι θα είναι καλή η συνεργασία μεταξύ μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι είναι καλή η βάση τη εργασία του εισηγητή και μετά από τι συζητήσει που ακούσαμε σήμερα το πρωί, προφανώ υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Καταρχά, είναι φατικό σημάδι το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διδαχθεί από τα ασφάλματα τη οικονομική κρίση και ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να συμπεριληφθεί και η κοινωνική διάσταση στη φάση κατάρτιση προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι πολλά εστραπολογίε κινούνται προ την κατεύθυνση αυτή και με χαρά θα τι υποστηρίξουμε. Είναι βασικό να κατευθυνθούν οι επενδύσεις και η ενίσχυση των κρατών μελών ε, από δημοσιονομικής άποψης, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο των περικοπών, των δημοσιονομικών, κοινωνικέ ε, κοινωνικές περιπτώσεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στους πολίτες. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ένας αντισταθμιστικός παράγοντας και χρονικά αλλά και χωρικά να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την τάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερασιμότητες, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερω προσεκτικοί. Κυρίως λόγω του αντικυκλικού χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά τον αντικτυπώ στους πιο ευάλωτους. Να δούμε επίσης τι μπορεί να γίνει με το follow-up σε ό,τι αφορά τις ε, συστάσεις αναχώρα και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αν υπάρχουν δηλαδή κράτη-μέλη τα οποία δεν ακολουθούν τις συστάσεις που τους έχουν χορηγηθεί, πού θα έχει αυτό αντίκτυπο στην ε, χρηματοδότηση που τους χορηγείται. Ενδεχομένω να χρειάζονται και άλλε δράσει, αλλά προφανώ και είμαστε ανοιχτοί για να αντιβρεθούν τα κριτήρια πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία περί ανεργία. Είναι αρκετά άκομψε αυτό το εργαλείο. Με χαρά λοιπόν να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να δούμε πού θα ενταχθεί και ο έλεγχος, ο κοινοβουλευτικός και η διαφάνεια. Αυτό προφανώς μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο κύριος ε, Λέιαρικ, ούτε ο κύριος Μαρτά είναι εδώ να δώσω το λόγο εν συντομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουμε καθυστερήσει κιόλα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Λίβια Γκάλμπο από την Καπαδελτά Εκφή. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο. Έτσι είναι γνωματότηση για την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων. Και εμείς ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για την πρόταση αυτή και να ακούσουμε την άποψή σα και να τη συζητήσουμε. Είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να επιταχύνουμε τι συζητήσει με το Συμβούλιο, που έχουν τελματώσει αυτή τη στιγμή, καθώ τα κράτη-μέλη περιμένουν ένα πολιτικό μήνυμα για το πώ θα προχωρήσουν με τι συζητήσει. Σε ό,τι φορά τώρα τι τροπολογίε που προτείνει ο εισηγητή, Θέλω να δώσω κάποιες περιττέρω εξηγήσει ε, για τα 30 δισεκατομμύρια για το κονδύλι αυτό. Διαβάσαμε τις τροπολογίες, την τροπολογία 25 και είμαστε θετικοί. Όμως ως Κομισιόν έχουμε το καθήκον προσεκτικά να εφαρμόσουμε τον προπολογισμό της Ένωσης και να ακολουθούμε το τι είναι διαθέσιμο στο μελλοντικό περιθώριο στον προπολογισμό. Γι' αυτό προτείνουμε να αυξηθεί το ανατοτόριο από την πρόταση του του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά αν αυτή η αύξηση δεν συνάδει με αύξηση στους ίδιου πόρου, τότε το διαθέσιμο περιθώριο θα είναι χαμηλότερο από το σημερινό. είναι αυτού. Επίσης, ε, το, το ποσό της υπεστήριξης ε, που θα δίνεται έχει επιλεχθεί έτσι ώστε τα 30 δισεκατομμύρια να αρκούν για να δοθεί υποστήριξη σε όλα τα κρατημέλη που στην τελευταία ε, οικονομική κρίση ε, πληρούν αυτό το μηχανισμό πυροδότησης και εμείς ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε το 10% των δημοσίων επενδύσεων πέρα από τα δάνεια που εγγυάται η πρόταση Προβλέπεται και δυνατότητα ο ESM, ο μηχανισμό σταθεροποίηση, να δώσει στήριξη σταθεροποίηση παράλληλα, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει την ικανότητα σταθεροποίηση τη λειτουργία. Όμω αυτό θα θα απαιτούσε συγγνώμη, την ανάπτυξη ενό συγκεκριμένου μηχανισμού στο πλαίσιο του ESM και τη συνθήκη του. Τροπολογία 26 τώρα. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την, ε, ε, γενικούς περιορισμούς που ε, παρέχονται από το Γενικό Κονδύλι. Θέλουμε να αποφύγουμε να είναι προσβάσιμη λειτουργία σε ένα ή μόνο δύο κράτη-μέλη. Γι' αυτό έχουμε βάλει το όριο ότι δεν θα πρέπει να υπερβάνουμε το 30% ε, του έκρεμους ποσού. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το όριο για να έχουμε ίσους κανόνες για όλα τα κρατη Και στην τροπολογία 28 πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ο κανονισμός να μην αμφισβητεί την ίδια του τη χρησιμότητα. Η τροπολογία φαίνεται να λέει ότι η ευρωπαϊκή λειτουργία δεν θα έχει αντίκτυπο στη σταθεροποίηση. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκ, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Η λειτουργία θα βοηθούσε να αποφευχθούν σπιράλ ύφεση όπου μειώνονται οι δημόσιες επενδύσεις και θα μπορούσαμε να αποφύγουμε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και επιπρόσθετα μέσω των δανείων θα μειωνόταν το μέσο κόστος του δανείου για ένα κρατός μέλος που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κλειδονισμό. Έτσι λοιπόν θα δίναμε ένα σημαντικό μήνυμα και θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των χρηματαγορών. Για την επιλεξιμότητα για τα 30 δισεκατομμύρια υπήρξε η ερώτηση τι εννοούσαμε με τον όρο αρχή. Εδώ εννοούμε ως το ποσό του δανείου όχι κάτι γενικότερο. Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ με τα κριτήρια. Να σχεδιάσουμε τη λειτουργία για να αποφύγουμε ηθική βλάβη και μόνιμες μεταφορές. Επικεντρώσαμε όμως τα κριτήρια στην συμπεριφορά των κυβερνήσεων. Δηλαδή, ένα κρατός μπορεί να έχει να ανοίξει μια διαδικασία όπως ε, ε, όμως δεν θα πρέπει να έχει αποφάση του Συμβουλίου που να λέει ότι το κράτος ε, δεν έχει λάβει διορθωτικές δράσεις για να βελτιώσει την κατάσταση. των αυτών, σημειώνουμε ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου και ανυπομονούμε για την ευκαιρία να συνεργαστούμε περαιτέρω μαζί σας για να βελτιώσουμε και το κείμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκτός αν θες να πεις κάτι πάρα πολύ σύντομα, γιατί μόλις μας μένουν 20 λεπτά για το τελευταίο σημείο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 12.30. Ερήκε. Μάλιστα. Ας ρηχτούμε στη δουλειά σα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλό το συμπέρασμα, θεωρώ, που μας δείχνει και τι πρόκειται να γίνει. Πάμε στο τελευταίο σημείο της τη διάταξη. θέσπιση του προγράμματο για τα δικαιώματα και τις αξίες. Η κυρία Λάμπερτ, είναι η συγγήτρια. Θα σα ζητήσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι για να μπορέσουμε να δώσουμε και το λόγο στους κοιόδης. Παρακαλώ. Δύο λεπτά να βρω τα χαρτιά μου. Here on the, uh, the establishment of the right. Εδώ έχουμε τη θέσπιση του προγράμματος για τα δικαιώματα και τις αξίες. Ουσιαστικά βλέπουμε μια συγχώνευση δύο εφιστάμενων προγραμμάτων. Εδώ έχουμε ένα ταμείο το οποίο θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα μέρη που είναι σχετικά με την απασχόληση. Αναφερόμαστε πάρα πολύ σε θέματα που αφορούν την εισαγωγή διακρίσεων στην εργαλεία και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι λοιπόν, εμεί ω Επιτροπή Απασχόληση θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα και να είμαστε σίγουροι ότι στο χώρο εργασία όλοι χαίρουν μια αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Αυτό ταιριάζει και με τη συζήτηση που είχαμε σήμερα για την έκθεση Κούκαν σε σχέση με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ένα από τα θέματα που θέλουμε να τονίσουμε, προσπαθώ να διατηρήσω όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες τις τροπολογίες, είναι να τονίσουμε την ανάγκη για την πρόθεση των δικαιωμάτων και των αξιών, όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών. Θα δείτε μια τροπολογία που εξετάζει το θέμα της συνεχιζόμενης χρηματοδότησης για το Equinet. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, δεδομένου ότι οι φορείς αυτοί υπάρχουν και έχουν συσταθεί για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφέρουν από του φορεί τη κοινωνία των πολιτών. Έτσι λοιπόν οι περισσότερε τροπολογίε που έχω καταθέσει έχουν να κάνουν και με τον τίτλο. Νομίζω ότι αυτό ανέκυψε και στη ΛΥΜΠΕ. Δηλαδή ε, πρέπει να μιλάμε για την ισότητα και τι αξίες για να είμαστε σίγουροι ότι προωθούμε και τη διάσταση τη ισότητας. Έχω τροπολογία 12 όπου μιλάμε εκεί ότι πρέπει να μιλάμε για ανθρώπους, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για πολίτες ε, μας ρωτάνε τι εννοούμε με τους πολίτες. Ε, χρησιμοποιούμε τον όρο με την ε, έννοια της συμπερίληψης ή μιλάμε για πολίτες με νομικούς όρους. Έτσι λοιπόν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε διατύπωση που να συμπεριλαμβάνει όλες τις ομάδες, να μην αποκλείουμε ομάδες από την πρόσβαση στο Ταμείο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες. Ε, μία ε, ουσιαστικά αναφέρεται στον ε, σύνδεσμο με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας ε, Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε εδώ καθώς ε, το σχετίζουμε αυτό και με το ρατσισμό online και με τη ρητορική μίσους. Ε, κάτι που προτείνω ακόμη έχει να κάνει με το παράρτημα, με τον ε, κατάλογο των δραστηριοτήτων να μπει στο διατακτικό. Υπάρχει δηλαδή, αυτό είναι τμήμα του κανονισμού και φυσικά υπάρχει πολύ ξεκαθαρά στο πεδίο εφαρμογής. Αυτά ήταν νομίζω τα κυρία σημεία που ήθελα να φέρω στην προσοχή σας και αναμένω και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστούμε. Μας μένει ακόμα ένα τέταρτο. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στους σκιώδεις συζητητές, αλλά θα τους παρακαλέσω να είναι πολύ σύντομοι, να μην ξεπεράσουν τα δύο λεπτά. Ο κύριος Κόζα, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Σα hogy ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί δεν έχω δύσκολο νόημα να σας ε, μεταφέρω. Η γνωμοδότηση αυτή θεωρούμε ότι αποτελεί εξαιρετική βάση για μια καλή ανταλλαγή απόψεων, για μια καλή συζήτηση. Οι τροπολογίε. δε θα μας απασχολήσουν, θα τις εξετάσουμε και θα είναι σίγουρα επικοδομητική η συνεργασία μας. Ένα θέμα θέλω να θέξω μόνο. Έχω την εντύπωση ότι όλες οι πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν να μπουν στο επίκεντρο τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι... έχει προσυπογράψει ε, στην ε, συνθήκη για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό που λείπει εδώ είναι το θέμα των μειονοτήτων. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να ενταχθεί κάπως καλύτερα. Και θα ήθελα να δείξω και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω και το εξή. Να επιδείξουμε προσοχή σε ό,τι αφορά τις εργασίες μας. Να μην αποταχθούμε προτάσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα δύσκολα θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Τέταρτο σημείο σε ό,τι αφορά τους δείκτες. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προκειμένου στην συνολική διαδικασία να τηρούνται συγκεκριμένοι δείκτες σε ό,τι αφορά τους πόρους και την ε, προσμέτρηση των πόρων. Χαίρομαι λοιπόν ε, και προσβλέπω στις μελλοντικές μας εργασίες. Είμαι αισιόδοξο ότι τελική ανάλυση θα προκύψει ένα πακέτο το οποίο θα ακολουθεί με σαφένεια τον δεδηλωμένο στόχο μας ε, για την παροχή βοήθειας προς τις οργανώσεις υποστήριξης του πολίτη και θα προωθήσουν και τις προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ζανάτο, και πάλι παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ με πάρα πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν ως τώρα και με τις περισσότερες τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Ως εκπρόσωπος των σοσιαλιστών και δημοκρατών θα προσπαθήσω να ενισχύσω περισσότερο την σχέση με τις τροπολογίες που θέλουν να τονίσουν την αναγκαιότητα να έχουμε ένα όσο πιο αποτελεσματικό μέσο που θα έχει θετικό αντίκτυπο κυρίως ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη συναγωγή διακρίσεων, τον κοινωνικό αποκλεισμό των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων. Θεωρώ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να μπορεί να προωθήσει τις κοινέ αξίες ε, στι οποίε βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί πολίτες θα πρέπει να ε, θεωρούνται ισότιμοι. Ε, όμως πολλές φορές βρίσκονται σε κίνδυνο. Ε, πολλές ε, φορές σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι ακροδεξιές απόψεις στην Ευρώπη, το πρόγραμμα Δικαιώματα για Αξίες πρέπει να ενισχυθεί. Με το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, ζητήσαμε από την Κομισιόν ένα μέσο που να μπορεί να υποστηρίξει τη δράση της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η απάντηση της Κομισιόν ήταν θετική, αλλά δεν είναι ακόμη επαρκής. Είναι όλο ένα και πιο δύσκολο για τις ΜΚΟ να εργαστούν και να συνσφέρουν στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μου, οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών δέχονται επίθεση και απονομοποιούνται και στιγματίζονται. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, ένα μεγάλο μέρο των κονδυλίων αυτών ε, πράγματι να πηγαίνει στις ΜΚΟ και μέσω ε, κάποιων πιο ευέλικτων οικονομικών μέσων σε ό,τι αφορά ε, τώρα το κονδύλι ε, για το πρόγραμμα αυτό. Λυπάμαι που δεν είχαμε μεγαλύτερη πρικοδότηση για ένα ταμείο που θέλει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα έτη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, το σχέδιο γνωμοδότηση. Συμφωνώ με την αναγκαιότητα οι δραστηριότητε ε, του προγράμματο ε, που βρίσκονται στο παραρτημένο να μπουν στο διατακτικό του κανονισμού και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων να έχουμε και το θέμα του βόκαση του advocacy. Ε, επίσης, ε, θεωρώ ότι ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του τίτλου του προγράμματος να προσθέσουμε την ισότητα. Ε, le Ευχαριστώ για τους στερετικούς και μεταρρυθμιστές. Σε Ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές, έχω να πω ότι τις παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή, τις εξέτασα ιδιαίτερως. Το θέμα λοιπόν είναι η προστασία της δημοκρατίας, της ισότητας, των μειονοτήτων και το καθεξής. Όλα αυτά προφανώς μας αφορούν όλους μας. Χαίρομαι που μετά από πολύ καιρό επιτέλους είδα μία πρόταση όπου και πάλι αναφέρεται η καλύτερη ενσωμάτωση των Ρωμά στην ε, κοινωνία. Ενδεχομένως να έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, και πεπιθήσεις ε, με την εισηγήτρια, αλλά το θέμα είναι στην επόμενη προγραμματική περίοδο να κοιτάξουμε και το θέμα των ομιλιών μίσους στο διαδίκτυο να κοιτάξουμε το θέμα των ατόμων με αναπηρία, κάποια θέματα που απτονται κάποιων θρησκευτικών ομάδων. Θα ήθελα ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα παιδιά και στα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, για το ίδιο. Ο κύριος Μαρινιάν Πιντό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια πολύ σύντομα για τη σημασία που έχει γνωμοδότηση αυτή για μένα σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση λόγω της ανόδου λαϊκισμών από δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι αυτή η έκθεση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για να οδηγήσει εκ νέου την Ένωση στις αξίες που είναι στην γέννησή της, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο να θέσουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ανησυχιών της. Μια πολιτική και οικονομική ένωση δεν μπορεί να έχει ελευθερία κυκλοφορίας μόνο ε, για ε, τα κεφάλαια και τα εμπορεύματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και για τους Ευρωπαίους. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά την άποψή μου ε, βρίσκεται στην πηγή της κρίσης και της θριάμβου ε, των αντιδραστικών δυνάμεων. Τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα έχουν γίνει σαν στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Έχουν μείνει στα λόγια, αλλά δεν ε, μπαίνουν στην πρακτική των ε, Ευρωπαίων πολιτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εκ ένα κεντρικό κεντρικό σημείο δράση για του πολιτικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι πολιτικέ. και να μην μείνει μόνο σε ωραία λόγια ε, τα οποία εκφωνούνται μόνο σε ορταστικέ περιστάσεις. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ δεν υπάρχει κάποιο, ούτε για το EFDD, ούτε για το ENF. Η κυρία Σιγήτρια λοιπόν ε, να δευτερολογήσει. Κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους για τα πολύ θετικά του σχόλια. Από ό,τι φαίνεται θα καταφέρουμε να εργαστούμε από κοινού για να βελτιώσουμε, ελπίζω, την πρόταση που έχει τεθεί επιτάπητος. Ε, καταγράφω αυτά που αναφέρθηκαν για συγκεκριμένα μέτρα σε τη φορά της μειονότητας, για παράδειγμα, και ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε τις κοινέ άξιες. Νομίζω ότι αυτό το συμμεριζόμαστε όλοι. Σε ό,τι φορά την προστασία δεδομένων. Θέλουμε ο κόσμος να κατανοεί και τα δικαιώματά του. Και για μας αυτό στην Επιτροπή απασχόληση, μας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα προστασία δεδομένων στον χώρο εργασίας. Δηλαδή και εκεί οι εργαζόμενοι να βλέπουν ότι δεν παρακολουθείται κάθε του κίνηση η κάθε φορά που πληκτρολογούν κάτι στο, στον υπολογιστή τους. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, συναδέλφους και θα περιμένω με ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ. Στις εβδομάδες 45-46 θα γίνουν συνεδριάσεις ε, των σκιωδών. 19-20 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί ε, και στην, εδώ στην Επιτροπή και, στην, και στις 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Επόμενη συνεδρίαση στις 18 Οκτωβρίου το πρωί, εδώ στις Βρυξέλλες. Ζητώ συγγνώμη που κάπως ε, σας πίεσα χρονικά στο τέλος. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς γιατί επιταχύναμε και άρα δυσκολεύσαμε και το δικό τους έργο. Καλό απόγευμα.